Eh, Περιμέναμε πολύ. Περιμέναμε ε, τους συναδέλφους να έρθουν. Η κυρία Μάρτσεν όμως ήταν εδώ στην ώρα τη, ήταν εδώ στι στις 3 και 3 λεπτά. Ε, περιμένουμε τόση ώρα, ή κάναμε υπομονή, αλλά Για κάποιο λόγο συνήθως ε, οι προνομιούχοι είναι καθυστερημένοι. Ε, εμείς σήμερα κάπου το κόψαμε στη μέση και ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Ε, έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε εδώ την πρέσβυρα την κυρία Μάρστεν. Να πούμε ότι ναι μεν θεωρίστηκε τον Αύγουστο και δεν ε, μπορέσαμε να τη συναντήσουμε πριν αναλάβει καθήκοντα, όπως ε, είχαμε προσπαθήσει και είχαμε συμφωνήσει με τη Βαρόνι Άστον. Αυτό γίνεται συνήθως. Η κυρία Μάρζον, όμως ε, είχε την ευγενή καλοσύνη και να της δώσω και συγχαρητήρια διότι ένα από τα πρώτα ραντεβού που είχε στο πρόγραμμά της ήταν να έρθει εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Θα συζητήσουμε την ε, πολιτική κατάσταση στο Σουδάν, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσπαθεί να βοηθήσει στη σταθερότητα και στην ε, πολιτική ελευθερία της χώρας. Υπάρχει μια παγκόσμια συμφωνία ειρήνης που αρχίζει να αποδίδει τους του καρπούς, αλλά ακόμα βέβαια έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας και υπάρχει και μια ε, σύμβαση και ένα δημοψήφισμα ε, το οποίο ε, θα γίνει για την ανεξαρτησία του Σουδάν, το οποίο φυσικά μπορεί να δώσει και ενδιαφέρουσες προπτικές στη χώρα, εάν είναι θετικό. Πριν δώσω το λόγο στην ε, κυρία Μάρστεν, ήθελα να υπενθυμίσω, αν και φαντάζομαι ότι ε, οι συνάδελφοι γνωρίζουν την ε, πρώτερη επαγγελματική σας εμπειρία. Είχατε μια πολύ καλή διπλωματική πορεία, ασχοληθήκατε πάντα με πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις διάφορες προηγούμενες αποστολές σας. Έχετε διατελέσει πρέσβυρα στο Σουδάν για τρία χρόνια και στο Αφγανιστάν και στην Ευρωγενική Επιτροπή στη Βασόρα, στο Ιράκ. Ε, πρόκειται για ε, θέσει θέσεις ε, και φυσικά είχατε και πάρα πολλά πράγματα να κάνετε εκεί. Θα ακούσουμε τώρα λίγα πράγματα και για την φοιτεία σας και για την ανάλυση που έχετε να μας κάνετε για το Σουδάν. Και αυτή η πρώτη συνάντηση μας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, το οποίο ελπίζω ότι θα είναι καρποφόρους για όλους μας και φυσικά όλοι έχουμε αυτές τις καλές προθέσεις. Να σας δώσω το λόγο και στη συνέχεια θα έχουμε συζήτηση και θα ακούσουμε τους συναδέλφους, ε, θα έχουμε πέντε ή έξι παρεμβάσεις για να μπορέσετε να απαντήσετε καλύτερα στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις που θα γίνουν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τον χαιρετισμό σας, αξιότιμα μέλη, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Όπως σας εξήγησε και ο Πρόεδρος, το Συμβούλιο με διόρισε κατόπιν πρόταση τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου τον Αύγουστο και ανέλαβα καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου, αντικαθιστώντα τον κύριο Τόρμπεν Μπρούλερ. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω στο Κοινοβούλιο σε αυτό το σύντομο διάστημα ε, μεταξύ του διορισμού μου και της ανάληψης καθηκόντων μου γιατί ήμασταν στις καλοκαιρινές διακοπές αλλά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην αρχή της θητείας μου. Συναντήθηκα με κάποιους από εσά άτυπα και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις προτάσεις σας και για τα όσα θα μου πείτε σήμερα και προσβλέπω σε τακτικέ συναντήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσά θέλουν να μεταβούν στο Σουδάν ή ε, έχετε κάποιο ενδιαφέρον για το Σουδάν. Ε, Σα παρακαλώ, μπορείτε να, κάλλιστα να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Ω ε, ειδική εκπρόσωπο ε, για το Σουδάν. Ε, έχω αναλάβει καθήκοντα εκ μέρου τη είπα τη εκπροσώπου της Κάθριν Άστον για να ασχοληθώ με θέματα ασφάλεια, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρωπιστική βοήθεια και οι επόμενοι μήνε θα είναι αποφασιστικοί για το μέλλον του Σουδάν. Το Σουδάν βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του, διότι βρισκόμαστε στο τελικό αποφασιστικό στάδιο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του 2005, που τελείωσε τον πιο μακροπνόθεσμο ε, μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο και έχουμε μία συμφωνία η οποία ήταν πολύ σημαντική για το μέλλον του Σουδάν. Η Συμφωνία Ειρήνης ε, περιλαμβάνει και ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Σουδάν και ένα ε, δημοψήφισμα για τη μελλοντική ε, κατάσταση στο Σουδάν, στο Νότιο Σουδάν, που θα γίνει το 2011. Από το δημοψήφισμα αυτό θα δούμε αν θα περάσουμε σε μια τελική πορεία ειρήνης και σταθερότητας. Από την ε, συνάντηση για το Σουδάν που έγινε στην Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία του πρώτου... Ε, αντιπροέδρου του Σάλβα και του Μαντάχα, ο οποίος ε, ε, είχε προσκληθεί από τον ε, πρόεδρο Ομπάμα μαζί με άλλους αρχηγούς κρατού και κυβερνήσεων και εκπροσώπους από περίπου 25 μέλη και οργανώσεις, κράτη-μέλη και οργανώσεις εμένα μου ζητήθηκε να βοηθήσω να προχωρήσουμε τις ε, στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αποφασίστηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 6 Ιουλίου Φέτο. και ε, τα συμπεράσματα αυτά συνοψίζονται σε μία ως εξής. Καταρχάς, να συνδράμουμε ενεργά στην έγκαιρη εφαρμογή της ε, Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας μαζί με την εφαρμογή αξιόπιστων δημοψηφισμάτων για το Νότιο Σουδάν ε, στις 9 Ιανουαρίου του 2011. Επίσης, να υποστηρίξουμε την δημιουργία θεσμών και να βοηθήσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια και ε, να ε, σεβαστούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Επίσης, να ενισχύσουμε την ασφάλεια και να καταλήξουμε σε μια ε, ειρηνευτική διαδικασία για την περιοχή του Νταρφούρ. Να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων και συνεργασίας με το Διεθνές ποινικό δικαστήριο και να διασφαλίσουμε και πρόσβαση σε όλο το Σουδάν. Ο ρόλος μου ως ειδική εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ε, και να υποστηρίξουμε για να έχουμε ένα ειρηνικό και σταθερό Σουδάν, αλλά φυσικά αυτό δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Θα πρέπει να είναι μια συλλογική προσπάθεια και στη προσπάθεια αυτή θα συνεργαστώ στενό με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ε, φυσικά και με τα κράτη-μέλη και επίσης ε, θα είμαι σε στενή επαφή με τα κόμματα στο Σουδάν, την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις καθώς επίσης και με διεθνείς εταίρους όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Έθνη και την Αφρικανική Ένωση. με τον ειδικό εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάλι Μανκέριος και τον κύριο Γκαμπάρη, με τον πρόεδρο Μπέκη και ε, το πάνελ εφαρμογής της Αφρικανικής Ένωσης και φυσικά και με άλλους ε, διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου θα ε, το περνώ επί τόπου ή ταξιδεύοντας στην περιοχή. Από τότε που ανέλαβα καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου, Έκανα μια επίσκεψη στο Σουδάν όπου συναντήθηκα με ανώτατους αξιωματούχους και πολιτικού και, ε, πολιτικούς ηθήνοντες στο Χαρτούμ και στη Τζούμπα. Και επίσης ε, ήμουν και στη Νέα Υόρκη όπως σας είπα ήδη για να ε, παραστώσει συνεδρίαση την περασμένη Παρασκευή και υπήρχαν και στο περιθώριο και άλλες συνεδριάσεις που αφορούσαν το Σουδάν. Έκανα συναντήσεις με τους Αμερικανούς, Κινέζους, Ρώσους, Βρετανούς εταίρους μου του ειδικούς εκπροσώπους για το ε, Σουδάν ε, στις χώρες αυτές και τις επόμενες εβδομάδες ε, θα επισκεφθώ και πάλι το Σουρά, στο Σουδάν για να συναντήσω ε, πολιτικούς εκπροσώπους στην Αφρικανική Ένωση και θα μεταβώ και στη Γενέβη. Πριν πω σε συγκεκριμένα στοιχεία της εντολής, επιτρέψτε μου να σας πω Δύο λόγια για την επίσκεψη ψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη την περασμένη Παρασκευή, στην οποία και παρευρέθη. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ψηλή η εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο. Η Βαρόνη Άστον και οι ψηλοί αξιωματούχοι από κράτη-μέλη συμμετείχαν. Έγινε επίσης μια προσπάθεια να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα. Δεν αντέχει το Σουδάν επιστροφή στη σύραξη. Θα πρέπει τα δημοψηφίσματα να γίνουν στην ώρα τους και να σταματήσει η βία και να επικρατήσει ειρήνη. Ο πρόεδρος Ομπάμα όρισε ε, την ε, το μέλλον του Σουδάν ότι θα πρέπει να είναι ε, ειρηνικό ε, σε συνεργασία με τα άλλα κράτη, αλλιώς θα υπάρξει απομόνωση. Και βεβαίως θα πρέπει να τιμωρηθούν οι, ε, οι πέτοι. Ο Αντιπρόεδρος Τάχα καλωσόρισε τα όσα είπε ο κύριος Ομπάμα και δήλωσε προθυμία να ανταποκριθεί το Σουδάν σε αυτό. Μίλησε για ένα νέο πνεύμα και ένα νέο δρόμο από την κυβέρνηση Ομπάμα που τελικά θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Ο Αντιπρόεδρος Σαλβακή ε, δήλωσε επίσης και τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει εγκαίρος το δημοψήφισμα γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση θα σήμαινε κίνδυνο επιστροφή στη βία. Πάντως ε, είναι πιθανό να επιλέξει την ανεξαρτησία το Νότιο ε, Σουδάν και ότι το Νότιο Σουδάν έχει κάνει προόδους την τελευταία πενταετία που δεν έκανε ολόκληρη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. θα πρέπει τα δημοψηφίσματα να γίνουν εγκαίρως και να γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, επιταχύνει και θέλει να επιταχύνει τις διαδικασίες. Για τον Ταρφούρη η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για την κατάσταση ασφαλείας και την ανθρωπιστική και καλεί όλα τα μέρη να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις στην Τόχα και ε, να υπάρχει πλήρης ε, πρόσβαση της UNAMID και των ειρηνευτικών στατευμάτων. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση επίσης θέλει ειρήνη, δικαιοσία και τερματισμό της ατιμορρησίας. Επίσης να ανανεωθεί η εντολή των ειδικών για ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι υποστηρίζει ισχυρά τη δέσμευση του Πρόεδρου Ομπάμα όπως και το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Έθνη και η Αφρικανική Ένωση και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Εμπέκη και η ομάδα του η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απευθύνει έκκληση στους Σουδανούς να αντιληφθούν τη μοναδική ευκαιρία που τους προσφέρεται. Νομίζω ότι ε, κατάφερε να συγκεντρώσει υψηλού επίπεδου διεθνή προσοχή σε μια κρίσιμη συγκυρία αυτή η συνεδρίαση. Ο Γενικός Γραμματέας ηγήθηκε τη συνεδρίαση, όπω και ο πρόεδρο Ομπάμα που αποφάσισε προσωπικά να παρευρεθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά εκπροσωπεί το και οι αντιπρόεδροι Τάχα και Σαλβακίερ άκουσαν τα μηνύματα ότι θα πρέπει να γίνουν εγκαίρω τα δημοψηφίσματα, να είναι δίκαια και ελεύθερα και αξιόπιστα και να γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι ευνοϊκή τώρα η συγκυρία γι' αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για τη δική μου εντολή, την κεντρική ιδέα και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει τους στόχους αυτούς. Σε ό,τι αφορά ε, τη συμφωνία τη συνολική για την ειρήνευση, ε, είμαστε μόλις 100 μέρες από το δημοψήφισμα για την αυτοδιάθεση του Νοτίου Σουδάν και το μελλοντικό καθεστώς ε, της περιφέρειας ABA. οι προετοιμασίε δεν πηγαίνουν όπω έχουν προβλεφθεί με του ρυθμού που θα πρέπει, ούτε η Εφορευτική Επιτροπή έχει οριστεί. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά να γίνει και δεν ε, υπάρχει χρόνο για χάσιμο. Η εγγραφή στου εκλογικού καταλόγου και η ψηφοφορία θα γίνει στο Νότιο Σουδάν, αλλά και σε τμήματα του, στο βορρά της χώρας που ζουν πολλοί ε, από το Νότιο Σουδάν και σε, στο εξωτερικό επίσης. Θα πρέπει, τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει ειρηνικά το δημοψήφισμα εγκαίρως και να αντανακλά ε, τις επιθυμίες ε, του λαού. Αυτό τονίστηκε στη Νέα Υόρκη επίσης. Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ε, φέρεται να έχει δηλώσει ότι στις 15 Νοεμβρίου θα αρχίσει η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Και επίσης φέρεται λοιπόν ότι στις 9 Ιανουαρίου ε, υπάρχει δυνατότητα να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για το δημοψήφισμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει, θέλει να στείλει ε, Επιτροπή Παρακολούθησης των Εκλογών για την προετοιμασία των εκλογών και θα είναι ορατή και πολύ ε, πολύτιμη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δίνει και τεχνική βοήθεια για την Εφορευτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος έχει στείλει τρεις εμπειρογνώμονε που συνεργάζονται, δύο στην Τζούμπα και ε, ένα είναι στην Χαρτούμ. Επίσης έχουμε ξεκαθαρίσει ότι τα διδάγματα που έχουμε βγάλει από την εκλογική διαδικασία, όπως αναφέρονται ε, στην έκθεση της αποστολής παρατήρησης των εκλογών, θα ληφθούν υπόψη στις προετοιμασίες ε, διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Ανεξαρτήτως ε, της ΑΝΜΙΣ ε, που είναι η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι θα στείλουν τον κύριο Αμκάπα και μια ομάδα και έχει ζητήσει από τις δύο πλευρές να δεχτούν για να ενισχυθεί η αξιοπιστία. Αυτό το πάνελ παρακολούθηση δεν θα είναι απλοί παρατηρητές εκλογών με την κλασική έννοια, αλλά θα έχουν μια επισκόπηση και των προετοιμασιών, καθώς επίσης και της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος και θα συλλέγουν πληροφορίες από όλες τις πλευρές συμπεριλαμβανομένων και προηγουμένων ε, αποστολών παρατήρησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις ρυθμίσεις μετά το δημοψήφισμα και τις διαπραγματεύσεις περί αυτού, θα έλεγα ότι στις διακομματικές διαπραγματεύσεις για τις ρυθμίσεις μετά το δημοψήφισμα έχει γίνει αρχή. Σε τέσσερις ομάδες εργασίας γίνονται συζητήσεις, καταλήγουν τα θέματα της οικονομικής, της χρηματοπιστωτικής κατάστασης, το χρέος, το νόμισμα, το πετρέλαιο, το νερό, οι διεθνείς συμβάσεις, τα θέματα ηθαγένειας κτλ. Συνεχίζονται οι εργασίες αλλά πρέπει να επισπευστούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτές οι υποδιαπραγμάτευση ρυθμίσεις ε, για μετά το δημοψήφισμα ε, να είναι συγκεκριμένες γιατί αφορούν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές και πιστεύω ότι για την ηθαγένεια και για το πετρέλαιο είμαστε κοντά ε, σε μια αίσια έκβαση της διαπραγμάτευσης. Ε, ανάμεσα στο βορρά και στο νότο λοιπόν θα υπάρξουν επικοδομητικές σχέσεις και θα υπάρξει διακομματική συνεργασία και πρέπει να μεριμνήσουμε να υπάρξει αυτή η διακομματική συνεργασία ανεξάρτητα από την έκβαση του δημοψηφίσματος. Αυτό είναι κυρία σημασία για το μέλλον του Σουδάν. Για το νότιο Σουδάν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ε, το κράτος του δικαίου την παροχή ελαχίστων υπηρεσιών και ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων στο Νότιο Σουδάν. Στι 17 ε, Σεπτεμβρίου ήμουνα σε μια τεχνική συνεδρίαση υψηλού επίπεδου στο Νότιο Σουδάν για την ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων. Ε, στεγάστηκε εδώ στα κτίρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με υποστήριξη του UNDP, του, ΟΗΕ δηλαδή, εδώ στι Βρυξέλλε και ο κύριο Ντέβιν Ντέγκ, ο Υπουργό Οικονομικών και Οικονομικού Σχεδιασμού, εκπροσώπησε το Σουδάν μα παρουσίασε ένα σχέδιο δράση που απαριθμεί 19 βασικές προτεραιότητες ε, για την ανοικοδόμηση των υποδομών της κυβέρνησης ε, μέχρι ε, να λήξει τον Ιανουάριο του 2011 μεταβατική περίοδο της συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας ανεξάρτητα από την έκβαση του δημοψηφίσματος οι δωρητές μεταξύ των οποίων και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησαν στην κυβέρνηση, ε, συνεχάρισαν την κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάνη για την βούληση αυτή να οικοδομήσουν την υποδομή και δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν ούτως ώστε να χτενίσουν αυτό το σχέδιο και ή δυνατόν να το υποστηρίξουν σε κάποια σημεία. Επίσης η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι θα κάνει και άλλη συνεδρίαση στην ε, Ουάσιγκτον στις 9 Οκτωβρίου αυτή τη φορά. Για τον Ταρφούρ τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ε, να συνεχίσει να εστιάσει τις προσπάθειές της στο Νταρφούρ γιατί η κατάσταση ασφαλείας και η ανθρωπιστική κατάσταση φυσικά δημιουργούν ακόμη ανησυχίες. Η βία στο Νταρφούρ έχει οδηγήσει σε θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, εκατομμύρια εκτοπιστέντες ε, που ε, ζουν ακόμη σε καταβλισμούς για πρόσφυγες του ΟΗΕ. Τους τελευταίους μήνες σημειώθηκαν και άλλα επεισόδια ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και στις παραστρατιωτικές ομάδες, σοβαρή βία ανάμεσα σε εθνοτικές ομάδες, επίσης βία κατά των ε, όσων εργάζονται για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, ε, κατά των πολιτών, ε, κατά των αξιωματούχων του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται στενά με την Αφρικανική Ένωση για τον Ταρφούρ και έχει δώσει σημαντική υλικοτεχνική και οικονομική στήριξη καθώς και προσωπικό στον Ταρφούρ από το 2004 μέχρι το 2007 και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν πάνω από 40% του κόστου της UNAMI δηλαδή τη κοινή ειρνευτική δύναμη του ΟΗΕ και τη Αφρικανική Ένωση. η βασική εντολή είναι η προστασία των αμάχων και φυσικά η παροχή ανθρωπιστική βοήθεια, βοηθώντα να δημιουργηθεί ένα ασφαλέ περιβάλλον. Από πολιτική πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση με συνέπεια έχει υποστηρίξει τι προσπάθειε ε, του ΟΗΕ, του κυρίου Βασιλέα, συγγνώμη, του κοινού δημοσιολαβητή ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει καλέσει όλα τα μέρη να συμμετάσχουν στις ε, ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Δόχα ε, και εκείνο διαβεβαίωσε ότι ε, θα απελευθερωθεί και ε, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις το Σεπτέμβριο στην Δόχα σχετικά με ένα Ισλαμικό κίνημα του Νότου του, Νοτιού Σουδάν. Ο στόχος είναι να καταλήξουν σε μια τελική ειρηνευτική συμφωνία και ο στόχος είναι όλες οι υπόλοιπε παραστρατιωτικές ομάδες, ο ε, ο στρατός του κυρίου Απελεγουάχη, του παραδείγματος χάρη, μεταξύ άλλων, ε, για να εισέλθουν ε, στις συνολικότερες προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη συλλογικά είναι από τους μεγαλύτερους ε, παρόχους ανθρωπιστικής βοήθειας ε, στο Σουδάν ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεχίζει να ασκεί σοβαρή πίεση για να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της ανθρωπιστικής βοήθειας. Γίνονται διάφορες επαφές σε μέρους περιοχές του Σουδάν και η Σουδανική κυβέρνηση εσχάτως υιοθέτησε και μια στρατηγική για τον Ταρφούρ συγκεκριμένα και μεταξύ των οποίων και η πρόθεση η επανεγκατάσταση των εκτοπιστέντων ε, και ε, το βασικό είναι τι σημαίνει επιτόπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκαθαρίσει ότι προτίθεται να εισέλθει σε διάλογο με την κυβέρνηση, ε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να υπάρχει αυστηρή συμμόρφωση με τις ανθρωπιστικές αρχές και σχετικά με την επιστροφή των εκτοπιστέντων στα σπίτια τους. Πρέπει να γίνεται με υποασφαλείς συνθήκες και να παρακολουθείται η επιστροφή της και φυσικά υπάρχει το θέμα Κατοχή κατοχής εδαφών που πρέπει να ρυθμιστεί. Ε, επίσης, ε, το Ανατολικό Σουδάν δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη σημασία του. Δηλαδή, οι χειρότεροι δείκτες ε, για το Σουδάν ε, είναι στην Ανατολή. Έχει προγραμματιστεί μία διεθνή διάσκεψη δωρητών και επενδυτών στο Κουβέιτ την 1η και 2η Δεκεμβρίου ο, ο στόχος αυτής της διάσκεψης όπου θα συμμετάσχει ένα ε, ε, ίδρυμα του Κουβέιτ, η Ισλαμική Τράπεζα, ε, το πρόγραμμα, το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ και η Σουδανική Κυβέρνηση. προετοιμάζεται τώρα λοιπόν η διάσκεψη και αναθεωρούνται όλα τα έγγραφα που θα συζητηθούν. Η κυβέρνηση του Σουδανέ έχει αναφέρει πως ευελπιστεί να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάσκεψη επενδυτών. Γνωρίζω ότι οι συνάδελφοί μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσουν το θέμα του Ανατολικού Σουδάνε γιατί θα πρέπει να προγραμματίσουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κοινοτικά κονδύλια για το ε, ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη του 2009 ε, και θα διοχετευτούν σε διάφορε επιμέρου περιοχέ ε, του Σουδάν, μεταξύ των οποίων και στον Ταρφού σε αυτέ τι τρει περιοχέ, αλλά και στο Ανατολικό ε, Σουδάν. Θα στραφώ τώρα στην συμφιλίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναλάβει δέσμευση να εργαστεί για τη δικαιοσύνη και την ασφαλεία για καταπολέμηση τη ατιμορρησία στο Σουδάν και συνεργασία με το Διεθνέ Δικαστήριο. Ο πρόεδρο Σεμπέκη είπε ότι χρειάζεται δικαιοσύνη ειρήνη και συμφιλίωση στην έκθεση που ε, εκπώνησε το πάνελ του ε, ε, επιφορτισμένο με τη μελέτη της κατάστασης του Ταρφούρ. Και προωθείται ο ρόλος λοιπόν του Διεθνούς Διαδικαστηρίου διότι λόγω της αμεροληψίας του και έχουμε υπενθυμίσει ότι υπάρχουν υποχρεώσεις σε βάση του καταστατικού της δρόμης ε, για όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Ε, τώρα, ε, στις 17 Σεπτεμβρίου, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας Justice Othman παρουσίασε την έκθεσή του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη και στις εισαγωγικές του παρατηρήσεις αναφέρει αυτός ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας. Αναγνωρίζει λοιπόν τη δέσμευση της Σουδανικής κυβέρνησης και τις θετικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί, αλλά τονίζει ότι σε άλλες ε, σε άλλου τομεί ε, δεν έχει σημειωθεί πρόοδο. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιτροπή παραδείγματο χάρη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ προβλέπεται αυτό στην ε, συνολική ειρηνευτική συμφωνία και άρα ελοχεύει κίνδυνο για το δημοψήφισμα και για την ασφάλεια των αμάχων μεταξύ άλλων. Τώρα, στο διάλογο που θα ακολούθησε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε το ζήτημα τη προστασία των αμάχων, των παιδιών στρατιωτών και των θεμάτων που σχετίζονται με την προετοιμασία διεξαγωγή του δημοψηφίσματο και τόνισε ότι χρειάζεται επέκταση της εντολής. Το ίδιο τόνισε, τόνισαν και οι ΙΠΑ. Πιστεύουμε ότι τι επόμενε ημέρε ε, θα γίνει ψηφοφορία για αυτό το ψήφισμα. Αξιότιμα μέλη, επιτρέψτε μου να σταματήσω εδώ. Ε, θα, ε, με μεγάλη χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας και θα ακούσω τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας σε αυτή την απαρχή της εντολής. Ε, της δυσχερέστατης αυτής της περίοδου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη να ξεκινήσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Μάρσδεν που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Οι ερωτήσεις μου αφορούν κυρίως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο μόλις αναφέρατε. Το ποινικό δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον ε, Ομάρ Αρμπασίρ και μετά από τα όσα έγιναν φέτος είπαν ότι η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι περιορισμένη αν μη τι άλλο και θα ήθελα να ξέρω εάν εσείς ε, αναλαμβάνοντας τα νέα σας καθήκοντα, σκοπεύετε να ενισχύσετε κάπως το ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε αυτή την περίπτωση. Το γεγονός ότι ο κύριος Αλμπασίρ εμφανίστηκε στην γένεια για το νεορτασμό του συντάγματος και δεν συνελήφθη, ε, είναι ανησυχητικό. Και επειδή έχουμε και την ε, Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής στη Λιβύη, το Νοέμβριο, φαντάζομαι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει και ο Μάραλ Μπασίρ. Εμεί θα είμαστε εκεί, θα έχουμε εκπροσώπηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών. Πώ θα συμπεριφερθούμε εμεί, εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Το πάνελ υψηλού επίπεδου για τον Ταρφούρ, το οποίο σύστησε η Αφρικανική Ένωση, έχει παρουσιάσει τα σχέδιά του για ε, μακροπρόθεσμη ειρήνευση στην περιοχή. Πώς μπορούμε όμως να βοηθήσουμε εμείς στην εφαρμογή των προτάσεων αυτών. Και η τελευταία μου ερώτηση. Να επανέλθω στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Με ανησυχεί το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μία επίσκεψη έκπληξη από τον Ομάρα Αλμπασίρ στη Λιβύη. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι αντίστοιχα φαινόμενα είχαμε στη Λισαβόνα πριν από ένα-δύο χρόνια. Βέβαια δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε την παρουσία του κ. Μπουκάμπα, αλλά ε, πραγματικά περιορίζεται η ελευθερία μας για να κάνουμε πραγματικές συζητήσεις πολιτικής ε, και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με αυτούς τους απαταιώνες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνο. Διαδικαστικό πρόεδρε μόνο. Σε δύο προηγούμενες ακροάσεις ανταλλαγές απόψεων είχαμε την εξής διαδικασία. Μιλούσαν οι συντονιστές ε, κατά σειρά μεγέθους ε, της ομάδας τους. Ξέρω ότι δεν είναι πολλά μέλη παρόντα, αλλά μου φαίνεται περίεργο. Πώς δώσατε το λόγο πρώτα σε ένα αναπληρωματικό μέλος μικρής ομάδας και όχι κανονικά ως ήθιστε πρώτα το ΕΛΚ, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι λοιπά όπως κάνουμε συνήθως. Ε, ε, πράγματι, ε, προσπάθησα να είμαι λίγο ρεαλιστέ. Τέσσερα άτομα έχω στον κατάλογο και πήγα να το δω χρονικά. Οι κυρία Αργεντίνη και εσεί ε, σηκώστε πρώτη το χέρι σα και ε, διάλεξα κάποιον χωρί να λάβω υπόψη μου αυτέ τι ε, ε προποθέσει. Οι συντονιστέ δεν ζήτησαν το λόγο, επομένω τίποτα. Είδα τον κατάλογο και διάλεξα. Κύριε Τάνοκ, θέλετε να παρέμβετε για κάτι άλλο ή μόνο για το διαδικαστικό. Υποθέτω ότι είμαι ο επόμενος ομιλητής ε, σε αυτή την περιπτώση. Πάντως μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, το ξέρω ότι έχουμε ε, ε λίγα μέλη. Μα είστε ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συγχαρητήρια, Ντέιμ Rosalind, για το διορισμό σας. έχουμε υπόψη μας και έχουμε συναντηθεί ότι έχετε πάρα πολύ αξιόλογη ε, σταδιοδρομία στο Foreign Office και διατελέσατε και ε, πρέσβη στην Χαρτούμ. Και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας είστε ε, ένας από τους υψηλόβαθμους διπλωμάτες εκεί και είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι απόψεις ε, βεβαίως είναι καυτή η καρέκλα σα και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ ε, για το Σουδάν το τελευταίο έτο. Είναι κρίσιμη χώρα, τεράστια, ε, τεράστια αποθέματα και κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και ε, ανθρωπιστική καταστροφή από το Ταρφούρ, τον Αφίλιο πόλεμο στον Νότο και επίσης τι γίνεται με ε, ένα πρόεδρο που είναι ο πρόεδρος Αλμπασίρ, ο οποίος ε, καταζητείται και θα πρέπει να προσαχθεί στο Διεθνές ε, Δικαστηρίο και διπλωματικά όλα αυτά πώς τα αντιμετωπίζετε. Έχω πάει και στο Νότο και ενδιαφέρομαι πολύ. Είχε έρθει εδώ αντιπρόεδρος του Νοτιού Σουντάν στην Επιτροπή μας. Μάλλον θα έρθει στο προσεχές μέλλον. Το είπατε στην εισαγωγή σας Ε, είναι ολιστηρό το έδαφος και μπορεί η Χαρτούμ να ε, το κάνει πιο ολιστηρός. Τι θα γίνει σε περίπτωση που το δημοψήφισμα δεν ε, μπλοκαριστεί για λόγους νομοθεσίας, διοικητικούς, γραφειοκρατικούς, αλλά λόγω νοθείας από το Βορρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει, θα αναγνωρίσει τον Νότο χωρίς δημοψήφισμα, με το Βορρά να μην υπογράφει τη συνολική ενευτική συμφωνία και να διώκεται κιόλας. Και τι γίνεται με τα τρια εκατομμύρια ε, νότιο Σουδανούς που ζουν στο βόρειο Σουδάν. Κινδυνεύουν. Θα τους αφαιρέσουν την ηθαγένεια, θα τους εκτοπίσουν, θα τους ε, εξορίσουν, θα είναι απάτριδες. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και για τον κύριο Ομπάμα που προσπαθεί να εξευμενήσει και το Βορρά και χαλαρώνει και, και αέρι και τις αμερικανικές κυρώσεις. Και ακριβώς επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείες εμφανίζουν μια αμφισημία απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και δεν έχουν ε, υπογράψει τη συνθήκη της ε, Ρώμης, το, τη συμφωνία της Ρώμης, ε, και μήπως οι Ηνωμένε Πολιτείες του υποσχεθούν ατιμορρησία και προστασία του κύριου Μπασί. Όχι ότι την αξίζει βέβαια, αλλά ε, για λόγους ε, ε, υποβοήθησης της διαδικασίας. Για την Κίνα είναι εύκολο να πείστε φαντάζομαι τους Κινέζους και τους Ρώσους και χώρες που έχουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τους Αμερικανούς, αλλά με τους Βρετανούς και τους Γάλλους τι γίνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Γιατί είναι τόσο ισχυρή η θέση σας έχει ανεξαρτησία το δικαστήριο, δεν θα δεχτεί παρεμβάσεις ε, στη δίωξη που έχει ασκήσει κατά του κυρίου Αλμπασίρ. Ε, και για την παρατήρηση των εκλογών, έχετε καμιά ιδέα ποιος θα είναι επικεφαλή και σε ό,τι αφορά το γραφείο σας, είναι αρκετά στελεχωμένο σας αρκούν οι ανθρώπινοι πόροι και οι οικονομικοί πόροι για να κάνετε τη δουλειά σας σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλου, τους συμβούλους, τις μεταφορές, γιατί ξέρω ότι είναι σε κακή κατάσταση οι δρόμοι στο Σουδάν. Και ένα τελευταίο Έχετε ε, βρετανικό διπλωματικό διαβατήριο, σας έχει δώσει το Foreign Office, γιατί είστε πρώτη πρέσβή, γιατί σε πρέσβης θα δίνουμε, σε βουλευτές όχι, σε ευρωβουλευτές ε, και σε υπουργούς όχι. Εσείς πώς είστε, αφού είστε και Βρετανοί ειδικοί πρόσωπος και έχετε βρετανικό διπλωματικό διαβατήριο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Thank you, Ευχαριστώ, Δυστυχώ δεν μπορώ να συμμεριστώ τη χαρά του Βρετανού συναδέλφου μου γιατί κανένας ε, υποψήφιος από τη Σλοβενία δεν επελέγει ε, για τον πρώτο γύρο διπλωματών που θα στελεχώσουν τη δική μας την υπηρεσία. Και χαίρομαι πάντως ε, με την αξιολόγηση της πρέσβειας μας δεν... Το μόνο στοιχείο που θα μου έλειπε είναι μια πιο εμπεριστατωμένη ε, πολιτική ανάλυση. Τι αναμένεται ότι θα συμβεί, τι θα συμβεί ε, στις 9 Ιανουαρίου. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας. Εσχάτως ε, συζητούσα με κάποιο κάποια πολιτικά στελέχη στο Σουδάν που συμμετείχαν και στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα και μου είπαν ότι αναμένουν εμφύλιο πόλεμο στις 9 Ιανουαρίου. Ε, ισχυρίζονται ότι ε, δεν ε, γίνεται να αποφευθεί ο εμφύλιος πόλεμος. Ποιο είναι το δικό σας σενάριο. Η συνεδρίαση της Νέας Υόρκης ε, οδήγησε σε κάποια σοβαρή αξιολόγηση του τι μέλη γενέστε ε, ανάλογα με την έκβαση του δημοψηφίσματος είτε είναι αρνητική είτε, είναι υπέρ του ναι είτε υπέρ του όχι. Ε, και επίσης μας είπατε ότι με την ιδιότητά σας μεταβήκατε στο Σουδάν και εγώ όταν την εποχή της μεγάλης κρίσης στον Ταρφούρ πήγα δύο-τρεις φορές στο Σουδάν ε, ξέρουμε προφανώς ε, πόσο αναξιόπιστη είναι οι πολιτικοί συνομιλητές μας ε, στο Σουδάν. Αναφερθήκατε σε κάποιους, Αμπτούλ Βαχίντ, παραδείγματος χάρη, και Καλίλ Ιμπραχήμ. Ε, όμως συνεχίζουν επικεφαλής. Ε, πολύ σημαντικών ε, ομάδων στο Σουδάν. Ε, δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνει ο διάλογος μαζί τους. Ο Καλίν, από όσο ξέρω, είναι στη φυλακή στη Γαλλία ή κάτι τέτοιο. Άρα δεν είναι η ορθότερη τακτική για να συνάψει κάποιος πολιτική συμφωνία με κάποιο άλλο μέρος. Διαβλέπω λοιπόν ε, ότι χρειάζεται σοβαρός διαλόγος με όλους επικεφαλής όλων των ε, ε, ενόπλων ομάδων ανταρτών, μιλώντας για τον Ταρφούρ, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Νότιο Σουδάν. Δεν είμαι πεπισμένος πως δεν ε, μίλησαν με πυγμή όλοι στη Νέα Υόρκη, στη συνεδρίαση που έγινε. Είναι τόσο σοβαρή κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω μετά την περιγραφή που μας κάνατε. Έχω σοβαρούς ενδιασμούς και πολύ φοβούμαι πώς θα αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα τους επόμενους μήνες. Πάντως, εγώ θα έρθω σε επαφή μαζί σας και κατά πάσα πιθανότητα θα πάω και εγώ ίδιο στο Σουδάν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φένσον τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρέσβυρα. Πολύ ενδιαφέρουσα και διεξοδική η ανάλυση σας. Είναι πραγματικά εξόχως ε, δυσχερής η κατάσταση ε, στο Σουδάν Έχουμε τα εισοδήματα από το πετρελαιό και τις πηγές του πετρελαίου που φυσικά έχουν τον σημαντικότερο ρόλο στη διαμάχη. Πρέπει να υπάρξει καταμερισμός ε, του εισοδήματος ε, από το πετρέλαιο. Ε, άρα υπάρχουν και ιδιωτικά συμφέροντα. Λογικό είναι. Αυτό μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε σχέση με τις προετοιμασίες του δημοψηφίσμα, σε σχέση με τη σταθερότητα της περιοχής, σε σχέση με το δημοψήφισμα, δηλαδή ακριβώς ε, ε, σε ποια θέση βρισκόμαστε σε σχέση με τα αλλοδαπά συμφέροντα. Ευχαριστούμε ε, κύριε Σφένσον. Κυρία Χάουταλα τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Μάστεν, είχα την τύχη ήδη να σας συναντήσω εχθές και Είμαι πεπισμένη ότι είσαι η σωστή ειδική εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σουδάν. Σας ευχαριστώ ε, για το χρόνο και την επίσκεψή σας. Σήμερα ε, ε, συναντήθηκα κάποιο από το γραφείο μου με τον Άλλη Αγκάμπ και τον Άπτελ Ομι Ακάκα που υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν που μας εξήγησαν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Σουδάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας, είπαν, μας μίλησαν για διώξεις, παρενοχλήσεις από τη τις ε, δυνάμεις ασφαλείας ε, και ότι αυτές οι ε, παρατυπίες είναι διαδεδομένες. Τι μπορεί να κάνει η αντιπροσωπεία της Ένωσης στη Χαρτούμ για αυτό το θέμα, πώς αντιλαμβάνομαι εγώ την κατάσταση. Θεωρώ ότι δεν έχει καταβληθεί πραγματική προσπάθεια για να συνεργαστούμε με τους ακτιβιστές και του τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς ως ειδική εκπρόσωπος μπορείτε να αναλάβετε δέσμευση βάσει της οποίας ε, θα εγκατασταθεί ένα ε, focal point, ένα σημείο εστίασης, ένα κοινό σημείο επαφής αν θέλετε στο Σουδάν ε, για να συντονίζει τη δράση όλων. Επίσης αυτό το σημείο επαφής μπορείτε να μεριμνήσετε ώστε να συνεργάσετε στενά με την κοινωνία των πολιτών στο Σουδάν, παραδείγματο χάρη, διοργανώνοντας ένα εργαστήριο για να συζητήσουμε ακριβώς πώς θα συνεργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών. Πάντως εγώ είμαι πεπισμένη ότι θα είναι κρίσιμη η συμβολή ε, των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων των σχετικών οργανώσεων στο Σουδάν. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ντεκάιζερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μάρτσεν, καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι επειδή σας γνωρίζω και σας έχω δει επί τόπου στη Χαρτούμ, χαίρομαι πάρα πολύ που ο δικός μας πρόσωπος εκεί είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει τόσο καλά την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο σας και νομίζω ότι ήταν καλή επιλογή ο διορισμός σας. Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε τις νέες σας εμπειρίες. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ξέρετε ότι σήμερα έχει διαδηλώσει το δρόμο στο οποίο συμμετέχουμε κι εμείς και ίσως να αναφερθήκατε στα θέματα για τα οποία έχω να σας ρωτήσω. Αν απαντήσατε ήδη, μην ξαναρχίζετε να απαντάτε, θα ρωτήσω τους συναδέλφους μου. Ε, το πρώτο, για το δημοψήφισμα, σίγουρα θα μιλήσατε, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης απόσχησης του Νοτίου Σουδάν όχι μόνο για την Αφρική αλλά για τον Ταρφούρ συγκεκριμένα. Θα είχε καμία επίπτωση αυτό, κατά την άποψή μου ναι. Γιατί έχουμε δει και εδώ εκπροσώπους του Νταρφούρ που δήλωσαν ότι ποτέ δεν θα ανεχόντουσαν κάτι τέτοιο. Μπορείτε να μας ε, διαφωτίσετε γι' αυτό. Το δεύτερο. Έγιναν εκλογές που δυστυχώς ε, χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη νοθεία με διαφορές στο βορρά και στο νότο. Και στο νότο οι ένοπλες δυνάμεις επενέβησαν με τρόπο πάρα πολύ δυσάρεστο και λυπηρό. Τι γίνεται εκεί, πώς ε, ακολουθούν, τι εξελίξεις ακολουθούν και το SPLE ε σε περίπτωση ε, δημοψηφίσματος τι δράση θα έχει η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό. Και στη συνέχεια, για τις εκλογές, η αντιπολίτευση στις προηγούμενες εκλογές ε, τις μποϊκόταρε και δεν εκπροσωπείται παρά μόνο πάρα πολύ λίγο στη διάφορα όργανα και στις συνελεύσεις και αυτές οι πρώτες εκλογές που υποτίθεται ότι ήταν μια μετάβαση προς ένα πιο δημοκρατικό καθεστώς και πιο πολυκομματικό στο Βορρά θεωρείται ότι υπάρχει οπισθοδρόμηση και από την άποψη αυτή οι εκλογές αυτές ε, απέφυσαν εις βάρος της αντιπολίτευσης λόγω της τακτικής που κράτησε αποχής από τις εκλογές. Ευχαριστώ. να Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, από πλευρά μου να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Μάρστεν. Δεν σας γνώριζα πριν, αλλά είχα ακούσει για σας και για το βιογραφικό σας. Νομίζω ότι φαίνεστε ένα από τα πιο κατάλληλα άτομα για να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, κύριε Μπρόκ. Τρία θέματα θα ήθελα να θίξω. Εν μέρη τα έχουν θίξει και κάποιοι από τους προλαλήσαντες. Το θέμα των ε, πετρελαϊκών εταιριών στο Σουδάν. Ε, προσπαθούν κάποιες εταιρείες να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο, ιδιαίτερα στις ε, συνοριακές περιοχές μεταξύ Βορρά και Νότου. Εγώ είχα πάει στην περιοχή, αλλά πριν από 10 χρόνια με μια αυστριακή πετρελαϊκή εταιρεία που δεν δραστηριοποιείται πλέον στην περιοχή, το βασικό πρόβλημα με τις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες επιτόπου είναι ότι συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται σε διαφορετικό πλανήτη. Είμαι λίγο ομοί, αλλά ε, φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται σε ποια χώρα δραστηριοποιούνται και τι προβλήματα υπάρχουν. Τι μπορείτε να μας πείτε για τις επαφές ίσως ε, ε, που είχατε μαζί τους και τι ρόλο διαδραματίζουν στην ειρηνευτική διαδικασία και στη διαδικασία που έχουμε να εξελίξει για το δημοψήφισμα υπάρχει ως συζήτηση το θέμα της κατανομής των εσόδων από το πετρέλαιο μετά το δημοψήφισμα, πόσα ε, θα κατανέμετε και δεν ξέρω αν εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να συνδράμουμε και να υποστηρίξουμε την όλη διαδικασία επιτόπου. Δεύτερον, ε, το ανέφερε και άδελφος Χάιντι Χάουταλα, ε, οι μελλοντικέ σα επαφές με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως ε, στο Χαρτούμ αλλά και σε άλλα μέρη. Ε, είτε πρόκειται για οργανώσεις γυναικών, είτε πρόκειται για περιβαλλοντικές οργανώσεις που ε, υπάρχουν, είναι ελάχιστες, αλλά υπάρχουν. Ε, χρειάζονται και αυτέ υποστήριξη από πλευρά μα και ενδιαφέρον από πλευρά μα. Ε, έχετε πρόθεση να κάνετε κάτι, να προχωρήσετε σε επαφές μαζί τους και να τους εμπλέξετε στο έργο σας. Και το τρίτο θέμα είναι οι πρόσφυγες από τον Νότιο Σουδάν που ακόμα ζουν στο Βόρειο Σουδάν, είτε σε ε, στρατόπεδα είτε αλλού. Ε, γίνονται επιβάλλεται σαρία σε όλους, είτε είναι μουσουλμάνοι είτε όχι. Και υπάρχουν προβλήματα, για παράδειγμα, γυναίκες στους ε, που φέρνουν ε, ενοπνευματόδη και τα πουλούν και αυτό απαγορεύεται βάσει της σαρία και φυσικά φυλακίζονται. Πώς έχει η κατάσταση επιτόπου, είναι περίπου 3 εκατομμύρια οι νότιοι Σουδανοί, οι περισσότεροι από αυτούς είναι χριστιανοί, δεν είναι μουσουλμάνοι και υπόκεινται στο νόμο της Σαρία που κάνουν, ενώ κάνουν κάτι που σύμφωνα με τη δική τους την ε, θρησκευτική επίστη είναι σωστό αλλά βάσει της Σαρία δεν ισχύει. Ευχαριστώ την κυρία Λούνετσι και έχετε ένα μακροσκελέστατο κατάλογο ερωτήσεων. Ε, κυρία Μάρτιν, δεν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Καταρχάς η ερώτηση της κυρίας Αργεντίνη και το θέμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όπως σας είπα, για το θέμα αυτό το, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει συστηματικά το δικαστήριο και το έργο του δικαστηρίου και ε, έχει ζητήσει από το Σουδάν επανειλημμένως να συνεργαστεί με το δικαστήριο. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος, όπως γνωρίζετε, τους τελευταίους μήνες ε, εξέδωσε τουλάχιστον δύο δημόσιες δηλώσεις ε, για την επίσκεψή της στο Τσάντ και στην Κένια. Ε, συγγνώμη, την επίσκεψη του Πρόεδρου Αλμπασάρ στο τσάτ και στην Κένια και υπενθύμιζε στις χώρες αυτές τις νομικές τους διεθνείς υποχρεώσεις. Νομίζω ότι είναι σαφής η θέση μας από αυτού. Ε, άκουσα τι μας είπατε για την διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής ε, στα τέλη Νοεμβρίου. Γνωρίζω ότι υπάρχουν συζητήσει αυτή τη στιγμή με την αφρικανική πλευρά, αλλά δεν θα ήθελα να επισέλθω σε περαιτέρω προμέρειες από αυτού, διότι ε, καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείται. για το πάνελ ε, του Προέδρου Μπέκη και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για την εφαρμογή των προτάσεών του. ενθαρρύνουμε τον πρόεδρο και την ομάδα του να συνεχίσουν και ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τμήμα της έκθεσης που αναφέρεται στην ε, ε, δικαιοσύνη και στη συμφιλίωση. Η εντολή που δόθηκε από τον πρόεδρο του Μπέκη στην Αφρικανική Ένωση ε, νομίζω ότι στη συνέχεια διευρύνθηκε και εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το ρόλο που διαδραματίζει ο πρόεδρος Ουμπέκη σε όλη την ε, ε, περιοχή αλλά και στο Σουδάν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, δώσει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να υποστηρίξει τα όσα έχει κάνει για τα όσα θα γίνουν για παράδειγμα μετά από το δημοψήφισμα. Κύριε Τάνοκ, μου θέσατε μία από ερωτήσεις. Πρώτον, τι μπορεί να γίνει αν η κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν ε, ακολουθήσει μονομερή προσέγγιση, πώς θα ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε εικασίες για το τι μπορεί να συμβεί. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επισημάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το δημοψήφισμα να προχωρήσει βάσει των διατάξεων της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας και θέλουμε να γίνει εγκαίρος και ε, να, είναι και, ε, να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα θεωρείται αξιόπιστο. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να επιμένουμε στην πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του CPA. Τη συνολική ειρηνευτική συμφωνία, γιατί αυτό είναι ο καλύτερο δρόμο να ακολουθήσουμε. Τώρα, για το τι θα γίνει με του ε, νότιου Ιδανού που ζουν στο βορρά, και εδώ τίθεται ε, σοβαρό ερώτημα, γιατί φυσικά έχουμε και βορείου που ζουν στο νότο είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα που συζητούνται ω τμήμα των διαπραγματεύσεων για το τι θα γίνει μετά από το δημοψήφισμα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οτιδήποτε και αν συμβεί, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οι πολίτες να έχουν μία εξασφάλιση ότι δεν θα αποτελέσουν στόχο, δεν θα βρεθούν στο στόχαστρο από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία και για αυτό το θέμα μεταξύ άλλων, διότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά για το θέμα του δημοψηφίσματος. Επομένως πρέπει να υπάρχει και μια δέσμη λύσεων. Μου θέσετε και μια ερώτηση για το ενδεχόμενο αναπομπή τη ε, εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Το Συμβούλιο ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών έχει τη δυνατότητα να κάνει αναπομπή, νομίζω για ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα όμω δεν μπορεί να την αρνηθεί τελείω. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Η Αφρικανική Ένωση είχε και κάποιο ενδιαφέρον για αυτή την περίπτωση, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο αποτελεί ενδεχόμενο. Ε, όπως σας είπα όμως είναι μόνο θέμα αναπομπής. Δεν υπάρχει εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, να ακυρώσει το ένταλμα σύλληψη που έχει δώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για την ε, ταυτότητα του επικεφαλής ε, της του, των παρατηρητών των εκλογών, εξ όσων γνωρίζω. Όσον αφορά τώρα το δικό μου προσωπικό και τα θέματα επιμηλητία. ανέλαβα τη θέση αυτή σε μια χρονική συγκυρία κάπως μεταβατική. Η εξωτερική υπηρεσία είναι που ανάπτυξε αυτή τη στιγμή. Και προς το παρόν εξετάζω τη σύνθεση της ομόδας μου, επειδή ακριβώς είμαστε εν εξελίξη. Ε, η Βαρόνια Άστον είναι περισσότερο αρμόδια, αλλά στο μέλλον θα συνεργάζομαι στενά με το νέο Γενικό Διευθυντή για την Αφρική, όταν θα βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος και φυσικά την ομάδα του. Στόχος είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ομάδα η οποία ε, θα ασχολείται με τα θέματα αυτά και θα σωματεθεί στην εξωτερική υπηρεσία. Ε, όπως σας είπα, είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα πρέπει να δω και, ε, εγώ, αν αρκεί το προσωπικό που έχω για να υποστηρίξει τα καθήκοντα που μας ε, αναλογούν. Αυτή τη στιγμή έχω ένα λεσέ πασέ για να ταξιδεύω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. με ρωτήσατε και αν μπορώ να σας κάνω μια βαθύτερη πολιτική ανάλυση του τι μπορεί να γίνει μετά το διποψήφισμα. Μπορεί να υπάρξουν και επεισόδια βίας και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια νευρικότητα στη χώρα για το τι μελγενέστε. Γι' αυτό άλλωστε και πιέζουμε και όλα τα κόμματα, από όλες, από όλες, τις συγγνώμη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ό,τι και να συμβεί θα γίνει με ειρηνικό τρόπο. Και ένας από τους καλύτερους τρόπους να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο σύραξη είναι να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τις συζητήσεις ε, για τις διαπραγματεύσει ε, στη διαδικασία του δημοψηφίσματος ε, που θα συμπεριλαμβάνει και το θέμα της ασφάλειας. Όσα περισσότερα συμφωνηθούν εκ των προτέρων, τόσο μικρότερος κίνδυνος προβλημάτων ελοχεύει. Όσον αφορά τώρα το πιθανό αποτέλεσμα, αυτό είναι θέμα του λαού του Σουδάν. Αυτοί θα αποφασίσουν. Νομίζω ότι είναι γνωστό της πάσης ότι υπάρχουν ε, ε, ισχυρές αποσχιστικές τάσεις ε, στο Νότο, αλλά οποιαδήποτε εικασία και να κάνουμε για το αποτέλεσμα, απλώς εικασία είναι. Το συζητήσαμε και στη συνεδρίαση της Νέας Υόρκης για το πώς ε, βλέπει ο καθένας το αποτέλεσμα, αλλά το δημοψήφισμα θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα κατόφλι. Θα έχουν, πρέπει να υπάρχει ένα 60% ε, ψηφοφόρων για να θεωρείται έγκυρο το δημοψήφισμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και αυτό σημαντικός παράγοντας ε, για το αποτέλεσμα. Αναφερθήκατε στην ανάγκη διαλόγου με τον Καλή Λιμπραχήμ και τον, ε, και τον Ουαχίδ. Ε, σαφώς θέλουμε να ενταχθούν στην Ειρηνευτική Συμφωνία. Ο Αχίντ είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι και δεν νομίζω ότι να είναι και φυλακισμένος. Ζω και αρκετά άνετα εμείς και άλλοι διεθνεί εταίροι φυσικά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε τον ε, Ουαχίτ και τον Ιμπραχήμ να ενταχθούν στη διαδικασία. Ο Χαλίλ ε, Ιμπραχήμ είναι στη Λιβύη νομίζω και ό,τι μπορέσουν να κάνουν οι Λίβοι για να τον ενθαρρύνουν να πάει στην Τόχα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Ο κύριος Βένσον ρώτησε τι γίνεται με την ε, κατανομή των εσόδων από το πετρέλαιο μεταξύ Βορρά και Νότου και τι γίνεται με τα ξένα συμφέροντα εκεί. Φοβάμαι πως δεν έχω και πολλά πράγματα να σας πω, θα τη σημειώσω την ερώτηση. Προφανώς ε, ο Βορρά θα χάσει σημαντικό τμήμα των εσόδων από το πετρέλαιο εάν αποσχιστεί ο Νότος, αλλά φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται και από τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν. Πρόκειται για ένα θέμα υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο πλευρών και νομίζω ότι ε, κάποιος άλλος, ε, νομίζω η κυρία Λούνατσεκ ε, ρώτησε κάτι αντίστοιχο. Ο ρόλος των πετρελαϊκών εταιριών στη διαδικασία του δημοψηφίσματος και για το πώς θα πρέπει να κατανέμετε το, τα έσοδα από το πετρέλαιο. Δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα από αυτού. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Νορβηγία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, υποστηρίζει και τις δύο πλευρές και τις προετοιμάζει για τις διαπραγματεύσεις για το θέμα των ε, εισοδημάτων από το πετρέλαιο, πώς θα κατανέμονται και αν μπορούν να συνεργαστούν για το πετρέλαιο, ώστε να διασφαλίσει ότι τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι απαραίτητα για αυτές τις συζητήσεις ε, θα είναι διαθέσιμα και να έχουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Οι Νορβικοί νομίζω έχουν κάνει πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά επί του θέματος και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ε, να ενθαρρύνουμε τις δύο πλευρές, να προσπαθήσουν να επιταχύνουν τις συζητήσεις και να συμφωνήσουν τουλάχιστον επ' αυτού. Κατόπιν δύο μέλη, η κυρία Χάουταλα και κάποιος άλλος με ρώτησαν για τα θέματα των ε, ανθρωπιστικών δικαιωμάτων. Και η κυρία Λούνατσεκ έθεσε την ίδια ερώτηση για τις οργανώσεις γυναικών και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Να σας διαβεβαιώσω ότι σκοπεύω όσο καιρό θα είμαι σε αυτό το πόστο να έχω στενές επαφές με τις ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που διαστηριοποιούνται τοπικά ε, για τα θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης ε, έχει ε, ε, φέρει στην επιφάνεια και κάποιες ε, μεμονωμένες υποθέσεις παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων και στο συμβουλευτικό όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στο Χαρτούμ έχει και αυτή ένα ε, τμήμα που ασχολείται μόνο με τα ανθρωπιστικά δικαιώματα. Η κυρία Ντεκέιζερ με ρώτησε τις επιπτώσεις μιας πιθανής ε, απόσχησης ε, του Νοτιού Σιδάν για τον Ταρφούρ. Το μόνο που μπορώ να σας πω ε, είναι ότι τα κινήματα στον Ταρφούρ δεν έχουν ζητήσει ανεξαρτησία. Ε, για τον Ταρφούρ το βασικό είναι αν θα είναι δημιουργηθεί, αν θα διαμορφωθεί μια ενιαία περιοχή στον Ταρφούρ και ακόμη είναι ανεπίλητο το ζήτημα. Ε, είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων στην Τόχα και ένα μεγάλο ε, κομμάτι του Νταρφούρ και η κοινωνία των πολιτών συγκεκριμένα έχει εκφράσει ένα ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ε, ε, περιφέρειας. Κοιτάξτε, οτιδήποτε συμβεί στις σχέσεις βορρά-νότου σίγουρα θα επηρεάσει και την κατάσταση στο Νταρφούρ. Αλλά δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, να πω ειδικότερα τι θα συμβεί για την αποστολή παρατηρητών του ΟΗΕ θα σας πω το εξής. Ε, πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την ε, αποστολή που κάναμε για το δημοψήφισμα. Αυτό ε, κατάλαβα στην πρώτη επίσκεψη που έκανα σε αρχές Σεπτεμβρίου στο Σουδάν. Um, στην έκθεση που συνέταξε η αποστολή σας υπήρχαν σημαντικότατες και ευστοχότατες συστάσεις, κυρίως σε σχέση με το δημοψήφισμα και εμείς προσπαθήσαμε ε, να τα τραβήξουμε και την προσοχή της ε, ε, Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ούτως ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι οφείλουμε να αντλήσουμε τα διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες και να τα χρησιμοποιήσουμε με επικοδομητικό τρόπο, ούτως ώστε όλα αυτά να γίνουν προς όφελος της διαδικασίας διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Αυτή τη φορά θα έχει πολύ σημαντικό το Αυτή την πρόθεση έχει, δηλαδή ε, και στις 79 κομιτείες του Νοτίου Σουδάν θα στείλει... Ε, προσωπικό και προσπαθούμε να, ε, προσπαθούν να ε, εκπαιδεύσουν επίσης αστυνομικές δυνάμεις και στο Βορρέδιο στο Νότιο Σουδάν για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Γίνονται δηλαδή θετικά βήματα και όντως ε, έχουμε αντλήσει χρήσιμα διδάγματα από την προεκλογική διαδικασία σχετικά με την επίπτωση που θα έχει αυτή η διαδικασία στο γενικότερο πολιτικό τοπίο και στον εκδημοκρατισμό της χώρας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το κυβερνών κόμμα καλύπτει και το βορρά και το νότο. Έχει πάρα πολλές έδρες στη Βουλή. Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν ελάχιστες έδρες σε προηγούμενες θητείες. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν σεβαστές ε, οι βασικές ελευθερίες, ε, ελευθεροτυπία, ελευθερία του συνέρχεστε, όλες οι ε, βασικές ελευθερίες και αυτό διότι πρέπει να γίνει ε, ένα αξιόπιστο δημοψήφισμα και να υπάρχει κατάλληλη πολιτική ατμόσφαιρα. Είναι απαραίτητο να γίνουν σεβαστές οι βασικές ελευθερίες. Εμείς θα συνεχίσουμε να το τονίζουμε αυτό και θα συνεχίσουμε ε, να υποστηρίζουμε μια προϊόντα διαδικασία εκδημοκρατισμού ε, στο Σουδάν. Το τελευταίο τώρα σημείο νομίζω ήταν ε, ε, για τις θέσεις ε, στο Βόρειο Σουδάνη, η κυρία Λούνατσεκ. Πολύ καλό το ερώτημά σας. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα ε, σε διάφορες ε, περιοχές ε, για τους μη μουσουλμάνους, κυρίως ως προς το κράτος του δικαίου. Ποιο μέσο έχουμε στη διάθεσή μας, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Μη Μουσουλμάνων. Είναι μία από τις επιτροπές που συστάθηκαν δυνάμει της συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας και φυσικά έχει διεθνή υποστήριξη η δράση της και την αξίζει ε, είναι το προφανέστερο μέσο ε, που μπορούμε να μετέλθουμε για να μεριμνήσουμε ώστε ε, να αποδοθεί ιδιαίτερη βάση σε αυτές τις υποεπιτροπές που στάθηκαν βάσει της συνολικής Ερευνευτικής συμφωνίας. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Μάρτεν, Πολύ καρποφόρα η συνάντηση, ε, σαφής ένδειξη της διάθεσής σας για συνεργασία και φυσικά και το πάθος ε, με το οποίο διεξάγεται το έργο σας. Ξεκινάει λοιπόν μια νέα σχέση μεταξύ μας η οποία θα συνεχίσει στους επόμενους μήνες και ελπίζω ε, έχει σημασία και για σας το γεγονός ότι μας ενδιαφέρει το θέμα και θέλουμε να συνεργαστούμε. Είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη σταθερότητα σε μια μακρινή χώρα ε, η οποία όμως μας αφορά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Διακόπτουμε και θα συνεχίσουμε στις 4.30 για να ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση ε, Cyrus Bene, colleghi, se Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουν οι εργασίες μας. Έχουμε να ψηφίσουμε την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των κοινοτήτων. Νομίζω ότι ο κύριος Σάιρους Βόλσκι έχει ζητήσει να κάνει μία παρέμβαση πριν ψηφίσουμε αν όντω θέλετε να μιλήσετε, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που ε, κάνουμε μια απόπειρα να ψηφίσουμε. Από την προηγούμενη εβδομάδα ήτανε. Είπαμε να αφήσουμε μια εβδομάδα να περάσει να το συζητήσουμε με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Δεν ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια για λόγους ανεξαρτήτης ε, θελήσεώς μας. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής και τους και και ε, τους υπολείπους. Προσπάθησα όσο μπορούσα να συμπεριλάβω τις προτάσεις τους. Νομίζω ότι ο συμβασμός τελικά που πετύχαμε είναι αρκετά καλός. Σεβάστηκα τις επιθυμίες των περισσότερων συναδέλφων να δοθεί ειδική έμφαση σε τρεις άξονες ισορροπιών, ε, γεωγραφική ισορροπία, ισορροπία φύλου και θεσμική ισορροπία. Και επίσης να έχουμε ένα ισχυρό στοιχείο ε, κοινοτικό στην ε, υπηρεσία εξωτερική δράση και συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Το πιο δύσκολο και επίμαχο ήταν το θέμα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, της γεωγραφικής ε, ισορροπίας και αντιπροσωπευτικότητας. Ε, συμφωνήσαμε και αποφασίσαμε, αλλά και ψηφίσαμε τον Ιούλιο, στο σημείο 7, αιτιολογική σκέψη 7 του θετικού ψηφίσματος που έχει επισυναυθεί στην απόφαση του Συμβουλίου και αναφερόμαστε στο άρθρο 6.1.6 της απόφασης για τη ισορροπία και θα πρέπει τα μέτρα να είναι ανάλογα για εκείνα που ε, είχαν αποφασιστεί στις 4 πρώτου του 2004 για αντίστοιχο κανονισμό του Συμβουλίου. Λοιπόν, τον Ιούλιο ψηφίσαμε, προσπάθησα να παραμείνω πιστός ε, σε αυτό το ε, ψήφισμα του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της παραγράφου 7. και στην γνωμοδότησή μου έχω κάνει δύο τροπολογίες 23 και 29 ε, που είναι ταυτόσιμες. Οι δύο βασικές ομάδες ε, ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και κάποιοι άλλοι συμφωνούν. Στην τελευταία εκδοχή για να ανταποκριθώ σε κάποια σχόλια και σε κάποιες αφιβολίες. Αποδυνάμωσα λίγο τις τροπολογίες μου και ε, τη γεωγραφική, την περιόρισα ε, και έβαλα κάποιους ενδεικτικούς στόχους πρόσληψης. Δεν είναι ποσόστοση, είναι ενδεικτικοί στόχοι ε, πρόσληψης για προσανατολισμό και όχι ποσοστώσεις. Επίσης ήθελα πω στους αδέλφους ότι ψηφίστηκε Σήμερα το πρωί της Επιτροπής Προϋπολογισμών με τις δικές μας τροπολογίες 23 και 29 που ταυτίζονται με τη δική μου πρόταση και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Και αν συμφωνήσουν οι συνάδελφοι και οι δύο επιτροπές θα στείλουμε ε, το ίδιο μήνυμα στους συναδέλφους ε, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Αν έτσι λοιπόν ψηφίσουμε... Ε, θα είναι καλή η αφετηρία και ο συμβασμό για να διαβάσουμε, επαναλαμβάνω, την άποψή μα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Και όταν θα πάω στον τριμερή διάλογο τη Δευτέρα, θα ακούσω τι έχει να πει ο, κυ... ο κύριο Ραπκάη, ο οποίο μα έχει τονίσει και στο παρελθόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούν τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Εξωτερικών, που είναι βασική, που είναι κρίσιμη και ο καλύτερο γνώστη ε, του αντικειμένου για το οποίο συζητούμε. Διότι δεν είναι μόνο προσωπικό το θέμα, αλλά και εξωτερική πολιτική. Δεν ολοκληρώνεται βεβαίω εδώ η διαδικασία αυτή. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Μετά θα πάει στην νομική επιτροπή και στην Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι είναι καλή αφετηρία η θέση μου αυτή και σαφής και ε, αποτελεί καλή βάση για μελλοντική εργασία. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και υποβάλλω την πρότασή μου στην Επιτροπή μας και νομίζω ότι αντικατροπίζει το ύφο, το πνεύμα, το γράμμα, τις επιθυμίες και τις ιδέες όλων των συναδέλφων για την κοινή μας ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης, το διπλωματικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να δουν την πρότασή μου όσο γίνεται ευνοϊκότερα και να την υπερψηφίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάιρους Βόλσκι. έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριο Μπρόκ. Για ένα λεπτό μόνο, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Äh, Κύριε Πρόεδρε, ε, δύσκολο θα είναι να μιλήσω σε ένα λεπτό και να σας παρουσιάσω αυτά που θέλω. Θα προσπαθήσω. Την περασμένη φορά είχα ζητήσει αναβολή. Έκτοτε ε, εξελίχθηκαν κάπως τα πράγματα. Η κυρία Άστον εξήγησε τι έγινε με τους πρέσβεις και πρέπει να διαπιστώσουμε ότι κινήθηκαν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση και στην ισορροπία των φύλων και στην γεωγραφική ισορροπία και στα υπόλοιπα. Οπότε δεν έχουμε πολλά αρνητικά εδώ. Το άλλο, ε, σε ό,τι αφορά τις ηγετικές θέσεις, φαίνεται ότι λύνεται και αυτό και έχει αρχίσει να αποδίδει προσπαθία μας. Γι' αυτό έχει απόλυτο δίκιο ο Ζεφ Σάριος Βόλσκι ότι ε, όλα αυτά είναι μια ολόκληρη διαδικασία και μέχρι τις 6 Οκτωβρίου που θα αποφασίσει, η Νομική Επιτροπή θα υπάρξουν και άλλες επαφές και του εισηγητού του κύριου Ράπκαι. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Βόρσκι, να μην μιλάμε για ποσοστώσεις, αλλά για ενδεικτική ε, ε, οδηγίες για πρόσληψη. Είναι και αυτό ένα στάδιο της εξέλιξης προς ένα σωστό αποτέλεσμα για να ανταποκριθούμε ε, στις επιθυμίες μας ως προς την ισορροπία. Θέλω να θυμίσω κάτι για να μην το ξεχάσουμε. Αυτό που διαπραγματευτήκαμε στο παρελθόν και μια συνάδελφος και εγώ και είναι ισχύον δίκαιο ότι θα πρέπει η ισορροπία να είναι δεδομένη. Είναι ήδη σήμερα απόφαση και σε κανονισμό του Συμβουλίου. Και αν δεν ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα το 2013 να ε, γίνει μια ενδιάμεση αναθεώρηση και να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Θα δούμε αυτά που θα ψηφίσουμε σήμερα και θα φροντίσουμε να εφαρμοστούν και σύμφωνα με το ισχύον ε, πλαίσιο. Ωραία. Τελευταία παρέμβαση. Ο κύριος Λάζορφ, σας παρακαλώ, προσπαθήστε τουλάχιστον εσείς να μιλήσετε για ένα λεπτάκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, κύριος Λάμστορφ. Ο κύριος Άρης Βόσκι είπε ότι ήταν δύο μεγάλες ομάδες που συμφωνούν. Ναι, αλλά πρόκειται για τέσσερις ομάδες που συμφωνούν και ε, θεωρώ λυπηρό ότι όταν μιλάμε για ισορροπία και αναλογικότητα Έχουμε χάσει τελείως την αξιοκρατία. Τα προσόντα, την εμπειρία, όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο. Τώρα βλέπω και χαίρομαι ότι έχει βελτιωθεί λίγο, έχει αποδυναμωθεί αυτό με τις τροπολογίες του κυρίου Σάρις Βόλσκι. Στις παραγράφους που γίνεται λόγος για την περίφημη αρχή Κίνοκ, ε, ενδεικτική στόχη, indicative targets. Πρέπει να πω ότι και εμείς και η δική μου πολιτική ομάδα είμαστε υπέρ της ισορροπίας και της αλογικότητας και στα θεσμικά και στα θέματα φύλου και στα γεωγραφικά. Πλην όμως έχω μια τεχνική ερώτηση και προφορική τροπολογία. Υπάρχει μια νέα προφορική τροπολογία του εισηγητού μας που αναφέρεται στην τροπολογία 17. Αλλά η τροπολογία 17 είναι τμήμα ε, της συμβαστικής 1. Τώρα η νέα προφορική αναφέρεται και αυτή στην τροπολογία παριθμών τη συμβαστική. Δεν το καταλαβαίνω από τον κατάλογο ψηφοφορία και προτείνω την εξή προφορική τροπολογία για το Compromise 1. Έχουμε μια ε, συμβαστική από τη 17 και τη 38 τώρα του κ. Σαρισβόσκη και τη συναδέλφου πράγματος. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού στην πρώτη παράγραφο στο 12.1 για τις συνθήκες ε, απασχόλησης θα πρέπει να βάλουμε κανόνες έτσι ώστε οι υπάλληλοι και οι προσωρινοί υπάλληλοι να είναι ε, υψής της ε, ικανότητας και ακαιρεότητας και να προσλαμβάνονται με βάση γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και δεδομένη ισορροπία φύλου. Προφορική τώρα τροπολογία. Τι θα πει με βάση τη γεωγραφική εκπροσώπηση και να επιζητούμε και τα προσόντα. Όχι, βάσει προσόντων και να επιζητούμε γεωγραφική ισορροπία. Γι' αυτό κάνω την εξή προφορική τροπολογία. Λέει στα αγγλικά. Η απασχόληση θα πρέπει να προσανατολίζεται στο να εξασφαλίζει για τους θεσμούς τις υπηρεσίες υπαλλήλων προσωρινών και μονίμων ύψης της ε, ικανότητας προσόντων και ακαιρεότητας. Ε, προσπάθεια να πληρούνται και κριτήρια γεωγραφικής ισορροπίας και ισορροπίας φύλου. Παρακαλώ να προσθεθεί αυτό και να ψηφιστεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πέτερλε. Ζητώ συγγνώμη. Ε, σας παρακαλώ εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω εδώ συζήτηση τώρα. Άφησα τον εισηγητή και κάποιον από τους κοιόδης εισηγητής που θέλησε να πει ένα-δυο πράγματα να τα πούνε. Αλλά αν έχετε κάποιες ενστάσεις για τον κατάλογο ψηφοφορίας που δεν μας επιτρέπει να ψηφίσουμε σήμερα, θα πρέπει να αναβάλουμε την ε, ψηφοφορία. Αν έχετε δυσκολίες, και δεν μπορείτε να βρείτε τους προσανατολισμούς ψήφους στον κατάλογο, δεν είναι αυτή τη στιγμή, η στιγμή να το συζητήσουμε. Ακούμε τις απόψεις σας, αλλά σήμερα προβλέπετε η ψηφοφορία, όχι η συζήτηση επί του θέματος. Και επίσης, αν έχετε μια αντίρρηση για μία τροπολογία, και θέλετε να κάνετε προφορική τροπολογία στη συγκεκριμένη τροπολογία, μπορείτε να παρέμβετε πριν ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία και ακολουθούμε τη συνήθεια διαδικασία. Ποιο είναι υπέρ κατά τη ε, προφορική τροπολογία και ψηφίζουμε. Αυτό πρέπει να κάνω εγώ. Εγώ θα ήθελα τώρα να κλείσει η συζήτηση εδώ ε, να ακολουθήσουμε τους κανόνες, να ξεκινήσει η ψηφοφορία και όταν έχετε ένσταση πριν ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη ψηφοφορία, ε, τροπολογία, υψώνετε το χεράκι σας, ε, κάνετε την ε, προφορική σας τροπολογία, την εγκρίνουμε, την απορρίπτουμε και από εκεί και πέρα προχωράμε. Συγγνώμη, αλλά έτσι έχουν οι κανόνες, πρέπει να τους σεβόμαστε, ακόμα και αν υπάρχουν ενστάσεις. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία 13, υπέρ. κατά αποχές να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση ελπίζω στο μεταξύ να έχετε βάλει τις κάρτες σας ε, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 13 60 ψηφίσατε, πέρασε ψηφοφορίας, 46 υπέρ, 14 κατά. Abbiamo l'emendamento. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 με την προφορική τροπολογία της κυρίας του, κυρίου Λάμστροφ υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Ποιος είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Ποιος είναι κατά. Ποιος δεν είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Σε αυτή την περίπτωση, Αν 40 κατά πρέπει να υπάρχουν ε, για την προφορική τροπολογία, τώρα είναι πολύ λιγότεροι. 5-6 ε, άτομα όμως αρκούν για να ε, μην ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Επομένως, ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ για τη συμβαστική τροπολογία 1. Το συγγνώμη. Ο κύριος Λάμστορφ, πρόεδρε, είναι τεχνικής φύσεως αυτό το θέμα. Η προφορική τροπολογία του κυρίου Σάριος Βόλσκι αναφέρεται και στην τροπολογία παριθμών 17, αλλά και στη συμβιβαστική παριθμών 1. Αυτό ερώτω. Στο 13 η πρώτη ψηφοφορία που κάναμε λέει προφορική τροπολογία του εισηγητού καλύπτει τις τροπολογίες 4, 17 κλπ αλλά καλύπτει τη 17. Τώρα, ο συμβιβασμός υπαριθμών 1 καλύπτει και αυτό το 17. Και ρωτώ τον κύριο Σαρισβόλσκι, αυτό που έχει υποβάλει ως προφορική τροπολογία για το άρθρο 17 ισχύει και για τη συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Allora, onorevole, onorevole Cyrus forse lei... Κύριε Σάρβις Πόλκη, μήπως μπορείτε εσείς να μας δώσετε την απάντηση. Συμφωνείτε με την ένσταση του κυρίου Λάμστροφ. για το συνδυασμό της συμβαστικής τροπολογίας 1 με την τροπολογία 13 και την προφορική τροπολογία που περιλαμβάνει και το σημείο 17 που συμπεριλαμβάνεται στη συμβαστική τροπολογία 1. Ακούμε την απάντησή σας και μετά θα συνεχίσουμε. Αν καταλάβαμε καλά την πρόταση της προφορικής τροπολογίας του κ. Λάμπστορφ, Πρόκειται απλώς για αλλαγή στη ταξινόμηση των κριτηρίων. Βάζει πρώτη την υπόθεση των προσόντων και την αξιοκρατία και τη γεωγραφική κατανομή και η ισορροπία τη διατηρεί, αλλά σε πιο χαμηλή σειρά. Aggiungiamo al compromesso 1 il termine non solo geografico ma istituzionale. Va bene, ma allora la proposta di chiarimento. Η πρόταση διευκρίνηση που γίνεται είναι η εξή. Προστίθεται στη συμβαστική τροπολογία 1 ο όρο θεσμικό στην τρίτη σειρά από το τέλο. Και αυτό επιτρέπει να υπάρχει ένας, ε, μια συνάφεια μεταξύ του συμβιβασμού και της περιφορικής ε, τροπολογίας. Κύριε Λάμπστορφ, αυτό θέλετε καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τεχνικό το θέμα. Κατά πότο το θεσμικό ε, θα πρέπει να μπει στο συμβασμό υπαριθμών 1. Υποθέτω ότι το θέλει αυτό η συγητής. Μάλιστα. Η προφορική τροπολογία όμως λέει προσλαμβάνονται ε, επί τη βάση των ενώ ταυτόχρονα ε, αποσκοπούμε κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να ψηφίσουμε. Έχουμε τέσσερις παρεμβάσεις για το σημείο αυτό. Δεν συμφωνώ και πολύ δεν νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία τώρα, να καθίσουμε να συζητάμε στο συγκεκριμένο σημείο, στο κείμενο και να έχουμε τόσες πολλές παρεμβάσεις για ένα κατάλογο ψηφοφοριών που έχει ήδη παρουσιαστεί. Αν θέλετε να το διευκρινίσετε, μπορείτε κάλλιστα να το κάνετε, αλλά πρέπει να έχετε καθορίσει τις θέσεις σας πριν φτάσουμε εδώ. Ο εισηγητής καταρχάς. Really, Πρόεδρε, είχαμε μία επιπρόσθετη εβδομάδα στη διαθέσή μας, άρα μην περιπλέκουμε τα πράγματα. Για το τεχνικό ζήτημα θα απαντήσω καταφατικά. Ε, εγώ υπέβαλα προφορική τροπολογία για τις 4, 13, 49, 52 και 14. Ε, ε διότι ήθελα να βάλουμε αυτές τις τρεις ισορροπίες, γεωγραφική, θεσμική και γεν... γενική ισορροπία, για την ισότητα των δύο φύλων ε, και γι' αυτό ε, σε ολόκληρο το κείμενο. Γι' αυτό έκανα αυτή την προσθήκη. Αλλά δεν θέλω να αναδιατυπωθεί και να πούμε while striving, δηλαδή ε, αποδυναμώνουμε το αρχικό κείμενο. Δηλαδή, όπως έλεγα και πριν, εσείς θέλετε απλώς να μπει θεσμική πτυχή στην τρίτη σειρά από το τέλος ε, της ε, συμβαστικής τροπολογίας 1 και έτσι ε, δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε αντιφατικούς όρους. Έχουμε τέσσερις παρεμβάσεις. Τάνοκ, Πέτερλεκ, ο κύριος Τάνοκ πρώτα. Δεν συμφωνώ βέβαια να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ένα σχόλιο, συγγνώμη πρόεδρε, γιατί είμαι αγγλόφωνος. Αν αλλάξετε τη λέξη with και βάλετε off, είναι πιο κοντά στην αξιοκρατία. Εδώ λέμε για κάποιους που να έχουν υψηλά προσόντα, αλλά έχει τους καλύτερους, όχι τα υψηλότερα, όχι να επικρατήσει ο ικανότερος, ο πιο άριστος και ο πιο άξιος. Γιατί όλοι λένε ότι είναι αξιοκρατία. Όχι, θα πρέπει να βγάλουμε το off και να βάλουμε το with. Και άλλες επιπλοκές. κύριος Μπράτνερ έχει ζητήσει το λόγο. Νομίζω πριν από τους υπόλοιπους. Η κυρία Μπράτνερ. Very quick point. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Θέλω να διευκρινίσω την τροπολογία του κυρίου Λάμστορφ. Λέει ότι ε, προσλαμβάνονται λόγω της γεωγραφικής εκπροσωπευτικότητας ε, και θα πούμε μετά ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε την ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτό εννοούσατε. Ναι, αυτή είναι η διατύπωση. Και θέλουμε να προσθέσουμε και τον όρο θεσμικός, institutional. Νομίζω ότι φτάνει τώρα, έτσι, μπορούμε να ψηφίσουμε. Το δεχτήκατε το with, έτσι δεν είναι. <laughs> μπορούμε να ψηφίσουμε με τις διευκρινήσεις αυτές για τη συμβαστική τροπολογία 1. Ε, προτείνω να μην αλλάξουμε άλλο το κείμενο. Διότι... Ε, Τέλο πάντων, ψηφίσουμε γιατί δημιουργούμε ε, επιπλοκέ. Δηλαδή, πριν το gender, πριν τα δύο φύλλα, θα μιλήσουμε για τη θεσμική ισορροπία. Ναι, αυτό θα κάναμε, γι' αυτό και προσθέσαμε αυτό το επίθετο και τώρα θα ψηφίσουμε για τη συμβαστική ένα με αυτή την προστίκη. Υπέρ. Κοντράρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στο 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν σηκώνετε τα χεράκια σας και βλέπω τους συντονιστές μόνο για να ξέρω σας. Παρακαλώ βοηθήστε με να μην καθυστερούμε κι άλλο. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. 19. Για το 19. Τροπολογία 19, άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν και 62. 46 υπέρ, 16 κατά. Επιβεβαιώνω λοιπόν ότι δεν σηκώνετε τα χέρια σας. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, συγγνώμη, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 40, όχι, καταπίπτει. Τροπολογία 23 με την προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ. Κυρία Μπραντνερ, θέλετε να παρέμβετε. Παρακαλώ. Μάλιστα, για να μην περιπλακεί ε, περαιτέρω το θέμα, θα ζητώ μία διευκρίνηση και θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά. Θέλω να εξασφαλίσω ότι αυτό το ε, τροποποιηθέν άρθρο όντω σημαίνει ότι το πρώτο κριτήριο είναι τα προσόντα και μετά η αναφορά του κοινόκ. Για λόγους ε, στελέχους πρέπει να είμαστε συνέτοι, όπως λέει το κείμενο, και εγώ θέλω να είμαι σίγουρη ότι έτσι το ερμηνεύει το σώμα, ότι το πρώτο κριτήριο είναι τα προσόντα. Αν αυτό ισχύει, εγώ θα αποσύρω την προφορική μου τροπολογία. Ευχαριστώ. Μπορεί να απαντήσει ο εισηγητής. Παρακαλώ. Μόνο τα άτομα με τα ανάλογα προσόντα μπορούν να ε, μπουν στην ευρωπαϊκή διπλωματία. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ωραία, εντάξει, τότε αποσύρω την προφορική μου τροπολογία. Καλώς. Σα δίνω για άλλη μια φορά το λόγο, αλλά είναι η τελευταία φορά που σας επιτρέπω να παρέμβετε, γιατί επαναλαμβάνω ψηφίζουμε, δεν ε, συζητάμε. Μια τεχνική διευκρίνηση στην ε, βουλγαρική εκδοχή λέει 31 Δεκεμβρίου του 2010 υπεραισιόδοξο, το 2020 στη βουλγαρική εκδοχή και επίσης μιλάμε για προσόντα και δεξιότητες σε άλλο σημείο, επομένω δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε εδώ, είναι σαφής η τροπολογία. Ε, σας παρακαλώ να ψηφίσουμε. Ε, 2010 η απόφαση λέει 2010, θα μείνει 2010, είτε είναι αισιόδοξο είτε όχι, αυτό θα μείνει. Αν συμφωνείτε το ψηφίζετε, αν διαφωνείτε δεν το ψηφίζετε. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία για τις 42. Αυτή τη φορά βιάστηκα μάλλον. 63 ψηφίσαντες, 33 υπέρ, 29 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 αποσύρεται, 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 καλύπτεται από την 23. Α, συγγνώμη, πρέπει να την ψηφίσουμε. 29 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 48 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τηλογική σκέψη 1, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ με την προφορική τροπολογία κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ α συγγνώμη εκπίπτει γιατί ψηφίσαμε την τροπολογία 3 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά δεν είδα καλά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 5. ...62 ψηφίσαντες, 63 πέρασε ψηφοφορία, 47 υπέρ, 16 κατά, 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, με την προφορική τροπολογία, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 αποσύρεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για τη γνωμοδότηση ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 54 υπέρ, 3 ε, κατά, 6 εποχές Προσθέτουμε και την ε, ψήφο του κυρίου Μπρόκ υπέρ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη. Ε, ο κύριος Μάουρο είναι υπέρ, ο κύριος Νταφ κατά και ένας ακόμα είχε σηκώσει το χέρι του. Τον κύριο Μπρόκ τον έχω ε, πει ήδη. Ωραία, προσθέτουμε μία ψήφο υπέρ, μία ψήφο κατά και θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση. Κύριε Μπρόκ, παρακαλώ. Μια στιγμή ησυχία, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ να γραφεί στα πρακτικά ότι αυτά να ερμηνευτούν και με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Ζαρισβόλσκη και μετά από τα όσα είπε η κυρία Μπράντνερ, ότι αυτό δεν ερμηνεύεται ως ποσόστοση και προέχει η αξιοκρατία πριν από οποιαδήποτε ισορροπία. Πρώτα η αξιοκρατία και μετά το παραμικρό ε, ε, περί ισορροπιών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνη σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, θα σημειωθούν στα πρακτικά οι απόψεις. Κύριε Μπράτνε. Ευχαριστώ, κύριε Μπροκ. Ε, πραγματικά ελπίζω να ερμηνευτεί προς την κατεύθυνση αυτή γιατί έχω ακούσει ότι διαφοροποιούνται οι απόψεις, γι' αυτό εμείς ψηφίσαμε αποχή. Λυπάμαι που το είπατε τώρα στο τέλος, αν το είχατε πει προηγουμένως ε, θα είχε βοηθήσει περισσότερο. Υπάρχει κάτι άλλο, ε, σας έχει παθιάσει αυτή η έκθεση. Ε, Πέτερλε, παρακαλώ. Πρόεδρε, δεν ε, το λόγο νωρίτερα. Ε, υπερψήφισα τη συμβαστική 1, αυτό ήθελα να δηλώσω, διότι είμαι ε, ήμουν πεπισμένο ότι δεν θα αλλάζαμε τη διατύπωση για τη γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα, δηλαδή ότι θα παραμείνει αυτό το κριτήριο. Πρόεδρος, μάλιστα με αυτό ισχύει. Απλώς προσθέσαμε το επίθετο θεσμικό. Στο υπόλοιπο κείμενο παραμένει αναλύωτο. Ε, ναι, και εγώ σύντομα να πω ότι ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι να έχουν την ίδια αντίληψη με αυτό που είπε τώρα ο Έλμαρ Μπρόκ. Δηλαδή ότι θέλουμε τους καλύτερους για την ευρωπαϊκή εξωτερική δράση. Και όταν προσλαμβάνουμε τους αρίστους, από εκεί και πέρα θα κοιτάμε τα διαφορά κριτήρια γεωγραφικά, ε, φύλου και θεσμικά για την ισορροπία. Αγαπητέ Έλμαρ, συμφωνώ και με την κυρία Έλμαρ, δεν κατέστρεψα τίποτα. Ε, γιατί χωράει και άλλες ερμηνείες στο κείμενο αυτό. Και με τη μορφή που έχει τουλάχιστον δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ικανοποιημένοι. Θα προτιμούσαμε μια πιο ξεκάθαρη διατύπωση. Ελπίζω στην πράξη και στην πρόληψη ε, στην πρόσληψη συγγνώμη, να ε, προέχουν πάντα τα προσόντα και η αξιοκρατία και όχι οποιασδήποτε άλλες σκέψεις. Ευχαριστώ για την ε, ψηφοφορία. Α, υπάρχει και κάποιος άλλος. Ο κύριος Βόμποντας, ζητώ συγγνώμη σας ξέχασα. Ναι, σύντομα πρόεδρε και εγώ δύο σχόλια μόνο. Πρώτον, κατανοώ την ε, αναταραχή και τα όσα δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι και ο εισηγητής. Ε, αυτά όλα είναι ένα μήνυμα σαφές και προς την κυρία Άστον αυτό το θέμα να ληφθεί υπόψη περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Και η ισορροπία γεωγραφική και η ισορροπία των φύρων και η κοινοτική μέθοδος ε, από τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εμείς εδώ στην Ομίγυρη θα πρέπει ε, να καταλαβαίνουμε ότι προέχει η αξιοκρατία και όχι τα γεωγραφικά ή το φύλλο. Ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε και στα δύο και η κυρία Άστον και το Συμβούλιο θα πρέπει να καταλάβει ότι και τα δύο θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται σεβαστά. Ευχαριστώ. One Γνώμη να πω στους συναδέλφους ότι χρειαστήκαμε ποσοστώσεις γιατί δεν ε, ίσχυε αυτό το περί προσόντων. Δηλαδή αν το σέβονταν αυτό όλοι περί αξιοκρατίας τότε δεν χρειάζονται ποσοστώσεις ε, όταν δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα προσόντα, τότε ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε ισορροπία από όλε αυτέ τι πλευρέ και γι' αυτό χρειαζόμαστε ποσοστό. Αυτό είναι το θέμα. Όχι αν είμαστε υπέρ ή κατά τη αξιοκρατία, ε, αλλά ε, φυσικά είμαστε υπέρ ε, τη ενίσχυση τη αξιοκρατία, αλλά δεν έγινε αυτό και άρα πρέπει να διορθώσουμε το αποτέλεσμα αυτή τη ε, μακρόχρονη προσέγγιση. Και τέλο ο εισηγητή και μετά ε, πρέπει να συνεχίσουμε την ημερήσια διάταξη. Με τον κύριο Κλίνκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, φαίνεται σαφώς ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για αυτό το θέμα και ελπίζω ε, να τραβήξει την προσοχή όλων μας. Ε, συμφωνώ απολύτως με όλους όσους τόνισαν πόσο σημαντική είναι η αξιοκρατία αλλά είμαι αντίθετη, αντίθετος με όλους ε, τους ε, υπόλοιπους που δεν υποστηρίζουν τις διάφορες ισορροπίες μεταξύ των οποίων και η γεωγραφική ισορροπία. Ε, δεν χρειάζεται να υπερτονίσουμε αυτό το θέμα, γιατί έτσι είμαστε επιθετικοί προς τις νέες χώρες. Δηλαδή, τι υπονοούμε, ότι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα υποψήφια από αυτές τις χώρες. Αυτό είναι θεμελιωδώς λάθος. Είναι εσφαλμένο, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάκριση μέσα στην Επιτροπή ή μέσα στο Ευρωπαϊκό Εκνοβούλιο. Είναι προϋπόθεση το προσόν. Κανείς δεν πρέπει να είναι επιλέξιμος για καμία χειρεύουσα θέση. Αυτό είναι προφανές, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα το προσόν για να υπάρχει ανισορροπία. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται όλοι να έχουν από το Eton, από το Cambridge και το Oxford ε, ε, ε, πτυχίο για να καταλάβουν τη θέση. Ένα λεπτό, Πρόεδρε, θα τελειώσω. Ε, δεν είναι γεωγραφικό ουδέτερο το προσόν γιατί ε, εξαρτάται από την κατάσταση στα διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διπλωματικό σώμα που θα εκπροσωπεί τη μισή Ευρώπη και όχι ολόκληρη. Ευχαριστώ. Ε, Ωραία. Είναι εδώ ο Υπουργό Κλίντου. Κύριε Πρόεδρε, πρόσβαλε το Πανεπιστήμιο, πρέπει να απαντήσω. Ε, δεν θα ανοίξουμε και συζήτηση ναι. τώρα. Μπορείτε μέχρι την Ολομέλεια να του πείτε ό,τι θέλετε. Έχουμε γνωμοδότηση, τη, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή. Συνεχίζουμε λοιπόν με την μέση διάταξη να μπει ο Υφυπουργό, όποιος θέλει να μείνει μένει, όποιος θέλει να φύγει φύγει. Όποιο δεν ενδιαφέρεται λοιπόν για τίποτα άλλο εκτός τη ψηφοφορία μπορεί να φύγει από την αίθουσα. Ε, πρέπει να μπει αντιπροσωπεία της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Ε, ε, Καθίστε συναδελφοί σας παρακαλώ. Ε, θα πρέπει να φύγει στις 6 και 4 ο Υπουργό. Δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Καλαθερίζουμε λοιπόν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων Παύλο Κλίμκιν και τον πρόεδρο της Επιτροπής για την Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, τον κύριο Μπόρις Τάρατζουκ. Η συνάντηση αυτή καταδεικνύει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και την αντιπροσωπεία της οποίας προεδεύει ο κύριος Κόβαλ. Η Ουκρανία συμμετέχει στην πολιτική γειτονίας ε, εμείς πάντα θέλουμε να έχουμε μια πιο καλή και πιο στενή συνεργασία με την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαπραγματεύσεις είναι εν εξελίξη, η συμφωνία διασύνδεσης βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των εργασιών μας. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα λοιπόν να ακούσουμε και τη δική σας ε, πλευρά για την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, για τα προσκόμματα και τις ευκαιρίες που μας χωρίζουν μέχρι να καταλήξουμε στη σύναψη αυτής της τόσο σημαντικής συμφωνίας. Νομίζω ότι οι παριστάμενοι συνάδελφοι θα ήθελαν να γνωρίζουν ε, το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της κυβέρνησής σας. Υπάρχει ε, εδώ και ο συνάδελφος Ταραζούκ, οπότε θα ακούσουμε και ε, το Κοινοβούλιο αλλά και το εκτελεστικό όργανο. Στο Κοινοβούλιο να επενθυμίσουμε ότι η πλειοψηφία έχει αντιπολίτευση. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Να ευχα... Ε, καλωσορίσω και τον κύριο Λεόνιτ Κότζαρα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της ε, αποστολής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε χρόνο 10 λεπτά. Αν μπορέσετε να τηρήσετε και αυτό το χρονοδιάγραμμα για να κάνουμε μια καλύτερη συζήτηση, έχετε το λόγο. Uh, thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλμπερτίνη. κύριε κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά που αισθάνομαι σήμερα που έχω την ευκαιρία να μιλήσω ε, στα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Είναι σημαντικό για ε, εμένα ως ε, αντιπρόεδρος, ε, συγγνώμη, ε, Υφυπουργό Εξωτερικών ως επικεφαλής των ε, διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σύνδεσης, αλλά ε, και ε, υπό την ιδιότητα που είχα στην διπλωματική μου σταδιοδρομία να ασχολούμαι επί δεκαετία και πλέον με ευρωπαϊκά θέματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία και χαρά που αισθάνομαι που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διετέλεσε και παραμένει ως θεσμικό όργανο υποστηρικτής θερμός των ευρωπαϊκών προσδοκιών της Ουκρανίας. Χαίρο ιδιαίτερος, όπως και στο παρελθόν, για το ιδιαίτερο πνεύμα που διέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς τις ευρωπαϊκές μας φιλοδοξίες. Πράγμα που αντανακλάται σε πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το 2010 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα ψηφίσματα, εξαιρετικά θα τα χαρακτήριζα, τα ψηφίσματα και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου της 25ης ε, Φεβρουαρίου για την Ουκρανία ε, τονίζει τη δυνατότητα που έχουμε βάσει το άρθρο 41 της συνθήκης ως ευρωπαϊκό κράτος να ζητήσουμε την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης αποδεικνύει ότι κάνει πρόοδους για την απελευθέρωση ε, της θεώρησης διαβατηρίων, βεβαίως ε, με καθορισμό ε, καταλόγου σαφών κριτηρίων προς την κατεύθυνση αυτή και το στόχο αυτό σε μια σύντομη παρουσίαση θα ήθελα να σας πω ότι τώρα είναι ευνοϊκή η συγκυρία στις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να υποστηριχθεί και περαιτέρω και θα ήθελα να σας προτείνω τρόπους ε, υποστήριξης αυτής της συγκυρίας. Πρώτον, θα πρέπει να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για την Ουκρανία δεν είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής ή καλύτερα δεν είναι ζήτημα μόνο εξωτερικής πολιτικής. Είναι κυρίως ένα ζήτημα ε, διεξαγωγή σε του ε, προγράμματος εσωτερικών μεταρρυθμίσεων για να ε, ευθυγραμμιστούμε με τα κριτήρια που απαιτούνται για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βλέπω βασικές προτεραιότητες για το αμέσως προσεχές μέλλον, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, Κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η συμφωνία ε, σύνδεση. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια τέτοια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, η βάση είναι η πολιτική σύνδεση και η οικονομική ολοκλήρωση και για μας είναι προστιθέμενη αξία εδώ και κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι η πραγματική ολοκλήρωση θα πρέπει να βασίζεται σε πλήρη ευθυγράμμιση της κρανικής νομοθεσίας προς την ευρωπαϊκή. Και αυτό θα πρέπει να είναι κινητήρια δύναμη για περαιτέρω ολοκλήρωση, διότι η συμφωνία που σήμερα έχουμε εταιρική σχέση και ισχύει ακόμα, είναι βεβαίως μια συμφωνία που αφορά μόνο τη συνεργασία θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία, αλλά όσο και να βελτιωθεί παραμένει η συνεργασία απλή. Θα πρέπει να υπερβούμε τη συνεργασία και να περάσουμε στην ολοκλήρωση, στην ενσωμάτωση. Και ακριβώ εδώ έρχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εκπόνηση των μελλοντικών εργαλείων και για την Ουκρανία. Και θα παρακαλούσα να ε, ρίξουμε μια νέα ματιά στα ε, μέσα και εργαλεία που θα πρέπει να εφαρμοστούν για αποτελεσματική εφαρμογή της επόμενης συμφωνίας σύνδεσης. Και δεν μιλώ μόνο για τον όγκο των οικονομικών συναλλαγών, αλλά και το είδος ε, των μελλοντικών ε, συνεργασιών μας, και, μέσων και εργαλείων, που για μένα θα πρέπει να εστιάζουν στην προσέγγιση της νομοθεσίας μας αναπόσπαστο τμήμα της μελλοντική συμφωνίας θα πρέπει να είναι ενός νέου είδους συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, ε, ε, βαθιά και συνολική, που για μας είναι αυτό σταδιακή επέκταση των τεσσάρων ελευθεριών στην Ουκρανία. Όχι επιλεκτική λοιπόν ε, ενσωμάτωση και ένταξη σε ορισμένου τομείς για όλες τις ελευθερίες. Ε, μιλώ και είναι βασικό σημείο ε, στις διαπραγματεύσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη προτεραιότητα. Βεβαίως ο διάλογος για την κατάργηση υποχρέωση θεώρησης διαβατήριων και εδώ επιζητούμε ε, έγκριση ενός ειδικού εγγράφου προγράμματος δράσης με ε, συγκεκριμένους στόχους για την Ουκρανία έτσι ώστε να καταργηθεί η υποχρέωση θεώρησης ε, διαβατηρίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει να τονίσω εδώ ότι για μας αυτό που χρειάζεται είναι λιγότερη πολιτική και περισσότερος ρεαλισμός και περισσότερη τεχνική θεώρηση ε, του διαλόγου για τη βίζα. Ήδη είμαστε καθοδόν ε, ε, για να αλλάξουμε το σύστημα θεός διαβατήριων μετανάστευση. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Το ειδικό πρόγραμμα που έχουμε για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων ε, και ε, για την μετανάστευση και κάποια άλλα προαπαιτούμενα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας τις εξελίξεις ε, στο διάλογο για την κατάργηση της θεώρησης. Επιτρέψτε μου και πάλι να υπογραμμίσω ότι δεν είναι καθόλου πολιτική η απόφαση την οποία επιδιώκουμε στο παρόν στάδιο. Είναι ε, σαφείς μεταρρυθμίσεις ε, και συγκεκριμένες. Αλλά χρειαζόμαστε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη προτεραιότητα. Είναι η ε, ημερήσια διάταξη, η ατζέντα για την ε, σύνδεση. Είναι πραγματικά ένα καινοτόμο έγγραφο. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτυχίες θα έλεγα για το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Και είναι μοναδική πρέπει να σας πω αυτή η συμφωνία αυτή ε, Ουκρανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη αρχίσαμε να εφαρμόζουμε τα συμφωνηθέντα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μελλοντική, τη μελλοντική συμφωνία σύνδεσης. Και δεν το θεωρούμε ως ε, νομικά δεσμευτικό, αλλά ως πολιτική υποχρέωση. Ε, έχουμε εφαρμόσει ήδη τα στοιχεία της συμφωνίας πριν τη θυσία Τέταρτη προτεραιότητα και όλος ιδιαίτερη για μένα είναι η συνεργασία σε θέματα ενεργειακά. Η Ουκρανία από πλευράς της έχει ε, αποδείξει την ε, προθυμία της να συνεργαστεί περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις την περασμένη εβδομάδα ε, υπογράψαμε στα Σκόπια ένα πρωτόκολλο ενεργειακής συνεργασίας Αρκεί να σας αναφέρω το νόμο για τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου που εγγράφεται πλήρως στο πλαίσιο της οδηγίας ε, της κοινοτικής 55 του 2003 και έτσι προετοιμάζει το έδαφος για αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου στην Ουκρανία και περαιτέρω ε, ένταξη της αγοράς και της Ουκρανίας στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως ε, θα δημιουργήσουμε στην Ουκρανία ένα ε, περιβάλλον επενδυτικό φιλικό προς τις επενδύσεις και τελειώνοντας χωρίς αυτό να είναι λιγότερο σημαντικό, θέλω να τονίσω κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βεβαίως βασίζεται σε προτεραιότητες και επιτεύγματα που σας ανέφερα, αλλά η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε τελική ανάλυση είναι ένα θέμα αξιών. Είναι θέμα ευρωπαϊκής σκέψης, νοοτροπίας, ε, ταυτότητας ευρωπαϊκής σε τελική ανάλυση. Πριν από λίγα χρόνια ε, επί ένα χρόνο συζητούσα κάποιες διατάξεις ε, να συμφωνήσω για την Ουκρανία. Για μας όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και ιστορικά, πνευματικά, διανοητικά η Ουκρανία είναι Ευρώπη και η θέση της είναι στην Ευρώπη. Και εδώ προσβλέπουμε στην υποστήριξη πραγματικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε στενά για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας και θα χαρώ να προσπαθήσω να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο θέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό και τώρα να ζητήσω από τον κύριο Τάραζουκ αν ε, μπορέσετε να είσαστε κι εσείς ε, συνεπείς και να τηρήσετε τα χρονικά όρια θα σας ήμασταν ευγνώμονες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα βάλω τα δυνατά μου ε, για να μην υπερβώ και το χρόνο μου όπως η Υφυπουργός Πλίνκιν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, όλα τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς ε, και όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Βλέπω οικία πρόσωπα, φίλους που εδώ και χρόνια εργάζονται για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της έκοινη γνώμης ε, των ε, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, το, για την Ουκρανία, για την προσχώρηση της Ουκρανίας. Ε, εδώ και χρόνια ασχολούμαι με το θέμα της συνεργασίας Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσα να σας πω το εξής. Έχουν υποθεί πολλά για τα πέντε περασμένα χρόνια και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι επειδή τα χαρακτήρισαν όλοι έτη έλλειψη σταθερότητας ε, στην Ουκρανία, θα ήθελα παρόλα αυτά να σας πω ότι καταλήξαμε σε πολύ σημαντικές συμφωνίες. Μεταξύ άλλων αρχίσαμε διαπραγματεύσεις για ένα νέο, μια συμφωνία πλαίσιο για ζώνη ε, ελευθέρου εμπορίου, και ολοκληρώνουμε τις διαπραγματεύσεις και θα τεθούν σε ισχύ δύο βασικές συμφωνίες για τις θεωρήσεις και για την επανεισδοχή. Επίσης άρχισε το καθεστώς ε, με εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης. Καταλήξαμε σε συμφωνία για μια κοινή, για μια συνθήκη μιας ε, ε, ενεργειακής κοινότητας ε, ανάμεσα στην Ένωση και την Ουκρανία. Είχαμε τις προεδρικές εκλογές σχάτως και ανέλαβε, ανέλαβαν νέες αρχές, νέα νέος πρόεδρος από τα μηνύματα που έχουμε ακούσει από εσά, τι καταλαβαίνω. Επειδή είμαι πρόεδρος τη κοινοβουλευτική Επιτροπής για την προσχώρηση τη χώρα μου στην Ένωση, θα έλεγα ότι οι νέε αρχές ε, καταδεικνύουν ε, την ε, βούλησή τους να ακολουθήσουν την θετική τροχιά των προκατόχων τους. Οπότε σημειώθηκε πρόοδος ε, τους ε, τελευταίους ε, μήνες κατά την διαπραγμάτευση της νέας Συμφωνίας Σύνδεσης. Ελπίζουμε ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου θα εισακουστεί και από τα λοιπά θεσμικά όργανα της Ένωσης, διότι δυστυχώς οφείλω να ομολογήσω πως οι διατάξεις ε, του ψηφίσματος, κυρίως σε σχέση με το ενδεχόμενο προσχώρηση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εισακούνται, δεν λαμβάνονται υπόψη από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Για την ε, ζώνη ελευθέρου εμπορίου, ε, ακούσαμε λίγα επικριτικά σχόλια κατά της αντιπροσ... ουκρανικής αντιπροσωπείας. Εγώ είμαι βουλευτής ε, στην Εθνοσυνέλευσή μας και φυσικά δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτήν την ε, κριτική κατά της ε, Ουκρανικής πλευράς. Ε, εφιστώ την προσοχή στο εξή. Εάν μιλάτε για ζώνη ελευθέρου εμπορίου ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να είναι ισότιμο εταίρο η Ουκρανία. Όχι μια επιπρόσθετη αγορά για τι ε, επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή λοιπόν την ε, σκοπιά θα έλεγα ότι θα πρέπει να αναζητηθεί συμβαστική λύση και από τι δύο πλευρέ όμω. Ε, και ένα, μια πραγματική συμβαστική λύση ε, ε, και να μην προταθούν στην Ουκρανική πλευρά αυτές οι μίζερες, οι σεχνές ποσοστώσεις, κυρίως για τη γεωργική παραγωγή. Ως προς το διάλογο για τις θεωρήσεις, έχουμε παρεμφερείς απόψεις, όπως και οι πρόσωποι της νέας κυβέρνησης, θεωρούμε ότι η Ουκρανία έχει κάνει πολλά για να διευκολύνει τα ταξίδια των πολιτών της Ένωσης ε, προς την Ουκρανία. Να σας υπενθυμίσω ότι από το Μάιο του 2005 και μετά εγκαταλείψαμε κάθε απέτηση θεώρησης για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Έκτοτε ε, έχουμε τη συμφωνία, τέτοια ισχύ η συμφωνία για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και αυτό οδήγησε σε ε, σημαντική αύξηση του αριθμού των θεωρήσεων Προ προς Ουκρανούς ε, ε, υπηκόους. Ε, τώρα, Πολωνία, Σλοβακία, η Ουγγαρία, οι γειτονικέ μα χώρε εισήλθαν ε, στη ζώνη Σέγγεν και τότε βλέπουμε ότι διάφοροι Ουκρανοί που ταξιδεύουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα προ αυτέ τι χώρε που προανέφερα ε, έχουν μειωθεί στον αριθμό. Δηλαδή, ε, τι σημαίνει αυτό, ότι οι Ουκρανοί δεν επωφελούνται από τη σχέση που έχουμε φτιάξει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα θεωρήσεων. Ε, για την ε, διασυνοριακή μετακίνηση και τις σχετικές διατάξεις δεν έχουμε πάλι κερδίσει πολύ. Λοιπόν, ως πρόεδρος κοινοβουλευτική Επιτροπής θα σας έλεγα ότι η Εθνοσυνέλευσή μας μας είχε θέσει το εξή. να παρακολουθούμε πώς και οι δύο πλευρές εφαρμόζουν τη συμφωνία και καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι διάφορε χώρε Ευρωπαϊκής Ένωση δεν πληρούν τις απαιτήσει και τις δεσμεύσει του. Γι' αυτό το λόγο θα έλεγα ότι μαζί με τους συναδέλφους μας ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ε, αποδώσαμε τη δέωσα έμφαση στο θέμα αυτό και ε, στην επικείμενη συνεδρίαση της ε, μεικτής ε, συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στο Κίβο και στην Οδέσα, τον, στην, συγγνώμη, στην Οδυσσό, τον Νοέμβριο, θα συζητηθεί αυτό το θέμα και θα πρέπει να ε, τεθεί υπόψη είναι όλων των μέλων και του Κοινοβουλίου και της Ουκρανίας. Ε, ποιο πρέπει να είναι το συμπέρασμα. Για να μην υπάρξουν παρανοήσεις, για να μην υπάρξουν προβλήματα ε, σε σχέση με τη Συμφωνία Διευκόλυνσης των Θεωρήσεων θα πρέπει να λειτουργήσουμε βάσει του συστήματος, δηλαδή να μην υπάρχει υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκούς της Ουκρανίας. Αναμένουμε λοιπόν στην επικείμενη σύνοδο που θα γίνει στις 22 ε, Νοεμβρίου θα διαπιστώσουμε πώς ε, θα προταθεί στην Ουκρανία ένα σχέδιο δράσης ε, για το καθεστώς εξαίρεσης από την υποχρέωση θεώρησης ε, εκφράζω λοιπόν τη σοβαρή ανησυχία για τις φήμες που κυκλοφορούν, ε, ίσως και εδώ στο Κοινοβούλιο, ότι δηλαδή η Ρωσία θα πρέπει να ε, έχει αντίστοιχο καθεστώς, να της προταθεί αντίστοιχο καθεστώς, αν όχι νωρίτερα, τουλάχιστον ταυτόχρονα με την Ουκρανία. μα, είναι ανησυχητικό αυτό, γιατί με τη Ρωσία εμείς θα προτείναμε το αντίστοιχο σιπικός ένωσης πριν από πέντε χρόνια. Ελπίζω να ασφαλώ, ελπίζω να με βοηθήσει να, να διασκεδάσω αυτές τις ανησυχίες, τις ανησυχίες που μοιράζονται παρεμπιπτόντως πολλοί Ουκρανοί. Επίσης, Ε, έγινε ένα θετικό σχόλιο από την ε, νέα κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες ε, εισήγαγε πολύ σημαντικά νομοσχέδια η νέα κυβέρνηση και σχέδια διεθνών συμφωνιών χάρη στις οποίες θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις προτάσεις για το καθεστώς εξαίρεσης από τις θεωρήσεις. Ευελπιστώ η κυβέρνηση να εκπληρώσει υποχρεώσεις της ε, ταχύτατα. Επίσης, ε, κρεμούν ακόμη διάφορα ζητήματα. Ε, βέβαια, τα επεξεργάζεται η κυβέρνηση και όλοι, βάζουν τα, όλοι βάζουμε τα δυνατά μας για να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση και όχι να λογομαχούμε. Επίσης, ε, πρόσφατα ε, συνάψαμε και τη συμφωνία, όπως έλεγα, για την ενεργειακή κοινότητα και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας. Ε, κανένας δεν πρόκειται να μας εμποδίσει από το να υλοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και έτσι να έχουμε και χρόνο για τη συζήτηση. Πάντως, ε, φυστώ την προσοχή σας ε, στο ότι δεν μιλούσα με την ιδιότητα του μέλους αντιπολίτευσης της Ουκρανίας. Έχουμε διαφορετικές απόψεις σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασης ε, στην Ουκρανία, αλλά μπορώ να επανέλθω όταν θα έχετε θέσει και εσείς ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Κόβολο, ο οποίο είναι για με την Ουκρανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μας δώσετε την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση για την Ουκρανία, προκειμένου να μπορέσουμε να ακούσουμε τις απόψεις της νέας κυβέρνησης, του νέου κοινοβουλίου. Και εδώ έχουμε τον κύριο Τάρατσουκ από την αντιπολίτευση σήμερα. Ε, Ευχαριστώ και τους δύο κυρίους για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε εις βάθος. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος σήμερα και δεν θα μπορέσουμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Δεν θα κάνω ερωτήσεις λοιπόν, απλώς να πω ότι ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα στη διάρκεια της ε, κοινή κοινοβουλευτική ε, ε, διάσκεψης που θα γίνει στο Κίεβο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Ως προς το θέμα των θεωρήσεων, Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανέκυψε με τη νέα κυβέρνηση και τον νέο πρόεδρο. πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων, θεωρούν ότι αυτή είναι η σωστή άγουσα και έτσι θα φέρουμε και του Ουκρανού στην Ευρώπη. Ω τμήμα τη νέα ε, συμφωνία διασύνδεση θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τα θέματα των θεωρήσεων, αλλά οι θεωρήσει ε, έχουν και νομικέ πτυχέ και είναι ένα ε, επιπλέον βήμα προ την ολοκλήρωση. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον Υφυπουργό να μας πει λίγα περισσότερα πράγματα για τις νομικές αλλαγές που θα μας οδηγήσουν με, στην κατάργηση των θεωρήσεων στο μέλλον. Εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων των διαβατηρίων, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι θέμα απλώς πολιτικής βούλησης είναι θέμα ελέγχων στα σύνορα, ε, θέμα ασφαλείας. Τα γνωρίζετε και οι δύο πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Επομένως, χρειάζεται η δική σας υποστήριξη προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι Το θέμα αυτό στο οποίο υπήρξε μια προκαταρκτική συμφωνία θα μπορέσει να υλοποιηθεί και να γίνει πραγματικότητα, διότι θα αποτελέσει πραγματικά ένα βήμα προς την ένταξη της Ουκρανίας. Σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας θα συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Ετοιμάζουμε και σχετική διεξοδική έκθεση που θα αναφέρεται στο θέμα των θεωρήσεων και των μεταξύ μας σχέσεων και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό θα συνεισφέρει τα μάλα. Ήθελα επίσης να πω στον Υφυπουργό και στον κύριο Τάρασουκ και εδώ δεν μιλώ τόσο ως πρόεδρος της, Επιτρο... της αντιπροσωπείας. αλλά ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ότι υπάρχουν ε, κάποιες ε, διαφωνίες στην Ουκρανία, έχουν αλλάξει η σύνθεση κάποιων επιτροπών Υπάρχουν πολιτικές ε, διαφορές στα θέματα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζουμε, που θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Και μήπως θα μπορούσατε να ρίξετε λίγο φως στην υπόθεση εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, αυτό θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για την ε, συνάντησή μας στο Κίεβο. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι ερίζουν οι απόψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για το πώς θα πρέπει να συζητήσουμε ε, τα θέματα της μελλοντική σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωση-Ουκρανία. Ξέρετε ότι ερίζουν οι απόψει και για τη διεύρυνση εν γέννη. Εάν η Ουκρανική ελίτ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει διαφορετική άποψη για τα θέματα αυτά, θα θέλαμε να το γνωρίζουμε οι φίλοι της Ουκρανίας, αυτοί που ενδιαφέρονται για την Ουκρανία, ε, δεδομένου ότι συμβαίνουν και πάρα πολλά πράγματα στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας, ε, να σταθώ στην ενέργεια, στην ενεργειακή κρίση, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα ετοιμαζόμαστε και για την ε, κοινή κοινοβουλευτική διάσκεψη στο Κίεβο και θα θέλαμε να γνωρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν θα καθυστερήσω άλλο. Οι απεργοί μα έχουν αλλάξει ολονών τα σχέδια. Πολλοί από εμά ήθελαν να ταξιδέψουν σήμερα και θα πρέπει να φύγουν. Και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που μα έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Κιόβαλ. Κύριο Γκάλερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και αγαπητοί προσκεκλημένοι από την Ουκρανία, η σημερινή συζήτηση αποτελεί μια καλή ευκαιρία μεταξύ φίλων να μιλάμε με λόγια σταράτα. Είναι σημαντικά αυτά γιατί κάτι αλλάζει στη χώρα σας και όχι προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής νοοτροπίας ή των ευρωπαϊκών αξιών. Ορισμένοι το αναφέρουν αυτό ως πολιτική σταθερότητα, αλλά θυμόμαστε την πικρή γεύση των εμπειριών του παρελθόντος που συνδέεται με αυτό. Δημοκρατία, ε, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου μας βοήθησαν και μας να είμαστε επιτυχείς. Ε, ε, και εμείς μιλούμε για θεσμική σταθερότητα και όχι άλλου είδους πολιτική σταθερότητα, όχι κάθετη ε, οργάνωση ε, της εξουσίας, γιατί ποτέ αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοήθησε. Γι' αυτό θέλω μια, ζώσα, ε, μια σφίζουσα δημοκρατία και στην Ουκρανία. Θα ήθελα να πω πολλά μαζί σας σήμερα για τα θέματα της Βίζας, για τη Συμφωνία Σύνδεσης και για θέματα δημοκρατικά, αλλά η χώρα σας ε, μου είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν μπορούσα να μην σας τα πω και αυτά. Σας ερωτώ λοιπόν, πριν τις δημοτικές εκλογές κατέβηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν επέτρεπε την ίδρυση νέων κομμάτων ούτε συνασπισμούς κομμάτων. Ή μάλλον ε, δημιουργήθηκαν νέα κόμματα αλλά δεν τους άφησαν να συμμετέχουν επιτόπου στις εκλογές. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς ή όλο και περισσότερο ε, οι μυστικές υπηρεσίες επισκέπτονται καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφους και άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών απρόσκλητοι. Γιατί ιδρύονται κόμματα επιτόπου με ένα αντίστοιχο όνομα περίπου με το όνομα του κόμματος της αντιπολίτευσης για να δημιουργηθεί σύγχυση στους πολίτες, εκφοβισμός από την εφορία, από τις τοπικές αρχές. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Πού το πάτε. Πώς να τα πω τώρα. Πώς εξηγείτε, πώς να το χαρακτηρίσω. Τη σύγκρουση συμφερόντων επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών να κατέχει και το μεγαλύτερο όμιλο μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή, ο μεγιστάνας του τύπου τώρα έχει γίνει και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών ή το αντίστροφο, έγινε καναλάρχης ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Φαίνεται αυτή η το αντιστροφο εγινε αλαρχης ο αρχηγος των μυστικων υπηρεσιων φαινεται αυτη η πορεια να διώχνει τη χώρα σας από την Ευρώπη και ε, να μην την φαίνει κοντύτερα. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει δημοκρατία, ευημερία και σταθερότητα για τη χώρα μακροπρόθεσμα. Και εδώ χρειάζεται μια πολιτική που να μην στρέφεται Προ την Ευρώπη και να μην την πλησιάζει μόνο στα λόγια, αλλά και στην καθημερινότητα και στην πράξη και στο πετσί του να τον νιώθουν οι πολίτε Και όχι να ευνοούνται αυτέ οι τάσει που δυστυχώ σήμερα παρατηρούνται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τρία λεπτά ο κύριο Μπροκ. Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότερο από τον κύριο ε, Γκάλερ ε, διότι με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον Υπουργό και στον παλιό μου φίλο Μπόρις Τάρατσουκ και να τους πω ότι έχουν δίκιο για τις συγκεκριμένες σχέσεις που θα πρέπει να έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία και να προχωρήσουμε. Και βεβαίω η ζώνη ελευθερών συναλλαγών θα πρέπει να έχει πλεονεκτήματα και για τι δύο πλευρέ. Για να ευδοκιμήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι μια ε, αμοιβαία υποφελή κατάσταση, win-win όπω ονομάζεται, και πολιτικά και οικονομικά. Και ο στόχος αυτός θα πρέπει να είναι. Γιατί με τη ζώνη ελευθερών συναλλαγών και την ε, ανατολική γειτονία θέλουμε αυτό να είναι ένα πρώτο στάδιο και για πιο στενές ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη λύση τύπου Νορβηγίας και τα λοιπά. Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά και στο παρελθόν και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι Πολύ λογική, και οικονομική, κυρίω η πολιτική. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα τη θεώρηση διαβατηρίων. Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν ναι, υποστήριζε ότι η Βίζα θα πρέπει να απελευθερωθεί πιο ε, γρήγορα ε, την Ουκρανία από τους άλλους ε, μεγάλους γείτονες, για πολλούς λόγους και πάλι. Και εδώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνει όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ξέρετε και... κάπου είχε γίνει και λόγος για μια τελωνιακή ένωση με τη Ρωσία. Τι γίνεται το συνεχίζει αυτό το σχέδιο και πώς συνάδει η ελεύθερη συναλλαγή με την Ευρώπη με την τελωνιακή ένωση με τη Ρωσία. Θα με ενδιαφέρει να μάθω. Και επίσης σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Γκάλερ τώρα προηγουμένως. Οι δυσκολίες της αντιπολίτευσης να βρούνε μέσα ενημέρωσης που να μεταφέρουν τη γνώμη της και τις απόψεις της, όχι μόνο ε, για λόγους οικονομικούς ε, και για άλλους. Και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και αν αλλάζει συνέχεια ο εκλογικό νόμος για να βολεύει αυτούς που κυβερνάνε, ε, δεν γίνεται. Ιδρύονται μικρά κόμματα ε, επιτόπου για να μην ε, επιτρέπεται η συμμετοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ας πούμε, για να μπλοκάρουν την κυρία Τιμοσέγκο. Και όλος περίεργος η δικαιοσύνη έρχεται να τα δικαιώνει αυτά τα φαινόμενα. Και η δικαιοσύνη τελικά δεν είναι ανεξάρτητη εξουσία, αλλά είναι το μακρύ χέρι της διοίκησης. Και ακούω ότι θα ισχύσουν και έκτακτες ρυθμίσεις για τις περιφερειακές εκλογές στο Κίεβο, κέντρο εξουσίας. Ε, δεν ξέρω, με ανησυχούν αυτά και με εκνευρίζουν σιγά σιγά και με προβληματίζουν. Και προς τα πού το πάμε, σε πραγματική δημοκρατία, με ένα κράτος δικαίου ανεξάρτητο ή επιστρέφουμε σε παλιά μοντέλα εξουσίας που ήταν μάλλον αυταρχικά καθεστώτα και τα εργαλεία κράτου δικαίου είναι εργαλεία και μόνο χωρί καμία ισχύ και χωρί να συνιστούν αξίε του κράτου. Ευχαριστώ κύριε Σεβερίν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τους εκρανούς ε, φιλοξενουμένους μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που βάλατε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα, διότι πριν από κάποιους μήνες ε, ακούσαμε ότι υπάρχει μία κόποση στην Ουκρανία και αυτό θα ήταν ε, μια τυχής εξέλιξη. Ε, θα ήταν κρίμα να ξεχάσουμε την Ουκρανία. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την Ουκρανία γιατί είναι σημαντική εν γέννη η Ουκρανία. Δεν μπορούμε να λησμονήσουμε την Ουκρανία γιατί είναι σημαντική για μας. Από την ε, πλευρά της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού μας προγράμματος. Θα πρέπει λοιπόν για άλλη μια φορά σήμερα να επαναλάβουμε ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν είναι ολοκληρωμένο εάν δεν έχουμε την Ουκρανία. Σαφώς υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Είχαμε προσδοκίες στο παρελθόν, έχουμε προσδοκίες και σήμερα και φυσικά δεν μπορούμε να κρύψουμε το γεγονός ότι πολλές φορές αποδεικνύονται φρούδες ελπίδες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε βέβαια είναι πρώτον να μην προσπαθήσουμε να παρέμβουμε στα μικροπολιτικά της χώρας, στη μικροδιαχείριση, γιατί δεν είναι και η δουλειά μας αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να αποφύγουμε να πάρουμε θέση, είμαστε υπέρ της αντιπολίτευσης της κυβέρνησης, να σκεφτόμαστε τη χώρα ως σύνολο και ε, τρίτον, ή δυνατόν να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να γίνει καλύτερη από τα δικά μας κράτη-μέλη, διότι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην Ουκρανία είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ και εκεί στις χώρες μας. Ε, Υπάρχει και ορισμένες φορές μία ε, πρόκληση, μία τάση για ε, πολιτερχική συμπεριφορά. Δεν θα σταθώ σε αυτό, αλλά θα ήθελα να συνεργαστούμε κατά τρόπον ώστε Ε, να κάνουμε αυτό που μας έδειξαν σήμερα οι καλοί μου φίλοι. Ο κύριος Τάρασουκ εδώ σήμερα ε, μίλησε ως Ουκρανός και όχι ως μέλος της αντιπολίτευσης. Και νομίζω ότι έχει σίγουρα εύλογα ε, πολύ διαφορετικές απόψεις ε, ως μέλος της αντιπολίτευσης, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα ελάχιστο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Ουκρανίας, και το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου, θα ήθελα να ζητήσω από τα πολιτικά κόμματα στην Ουκρανία να συνεργαστούν για την προαγωγή αυτής της Ουκρανικής ατζέντα. Ε, ε, εντάξει, σαφώς θα αντιπαρατίθεται διότι είναι κυβέρνηση και αντιπολίτευση. αλλά νομίζω ότι πριν ε, ρωτήσουμε την Ουκρανία τι έχει να μας πει για την εξωτερική της πολιτική, θα πρέπει να αναρωτηθούμε εμείς τι στάση κρατάμε προς την Ουκρανία, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις εκεί. Και επίσης, μια ερώτηση προς ε, ε, τους δύο προσκεκλημένους μας πώς ε, αντιδράτε στην πρόσφατη δήλωση της κυρίας Άστον που λέει ότι η Ουκρανία δεν έχει ως στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι είναι σωστή η περιγραφή της κατάστασης ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σεβερίν. Ο κύριος Τάνοκ για τρία λεπτά. Η Βαρόνια τον έκανε λάθος. δεν άλλαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτική. Το ΝΑΤΟ το έκανε. Αν συμβεί αυτό, τι να πω, θα είμαι σε απόγνωση. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Συγχαρητήρια, γιατί σήμερα χθε ήταν και η εθνική σας εορτή. Ε, και, και το είδα όταν κοίταζα <laughs> την ατζέντα μου, γιατί έχω να πάω σε ένα πάρτι σήμερα το βράδυ. Ε, και δηλώνω ότι είμαι ε, πραγματικός φίλος ε, και εγώ και το κόμμα μου της Ουκρανίας παρότι δεν ασχολούμαι τόσο επισταμένα όπως το παρελθόν με την Ουκρανία αλλά πάντως συγχαρητήρια για τις προσπάθειές σας για τη Συμφωνία Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και τη διατλαντική συνεργασία όπως και ο συνάδελφος ο κύριος Μπρόκ θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να γίνει πρώτα με και μετά με τη Ρωσία συμφωνία και η Ρωσία έχει προβλήματα γιατί έχει την Απχαζία, ε, την Τρασνιστερία ε, και διάφορες άλλες εμπόλεμες ζώνες παγωμένες ε, και υπάρχει θέμα αναγνώρισης της ηθαγένειας των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτά τα εδάφη για να μην σας μιλήσω για το Βόρειο Κάφκασο και τη βία και την εγκληματικότητα εγώ πολύ ανησυχώ αν υπάρξει ολική εξαίρεση των θεωρήσεων για τη Ρωσία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχω και Τώρα θα βάλω το άλλο μου το καπέλο, γιατί είμαι και εισηγητής του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή αυτή για την προσχώρηση, ευελπιστώ, του Μαυροβουνίου, ε, μία μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χτες συνεδριάσαμε, είχαμε μεγάλη αντιπροσωπεία, πολλοί βουλευτές ε, και δεύτερη φορά επίσημα αναφέρθηκε το ότι στις διαπραγματεύσεις στις δικές τους για την προσχώρηση στον ΠΟΕ, γιατί αυτό είναι ένα από τα πρώτα κεφάλαια που πρέπει να κλείσουν για να είναι υποψήφιες στην Ένωση, πρέπει να είναι μέλη του ΠΟΕ, ε, ο, ε, ο, η Ουκρανία ε, μπλοκάρει την προσχώρηση λοιπόν του Μαυροβουνίου για λόγους που δεν πολύ καταλαβαίνουμε παραδείγματος χάρη πρόσβαση στις αγορές Σερβίας δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο ποιος είναι ο πραγματικός λόγος διαφωτίστε με Υπουργέ αλλά πάντω το συζήτησαμε με, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τον Επίτροπο Φίλε, κατηδίαν. Θα ε, ε, συνεχίσω να ε, επιμένω. Θέλω να μάθω γιατί εσεί παρεμποδίζετε την προσχώρηση του Μαυροβονίου στον ΠΟΕ, γιατί σχεδόν καθόλου εμπορικέ συναλλαγέ δεν έχετε. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Ποιο είναι το κίνητρο τη κυβέρνησή σα για να τηρεί τέτοια στάση και ήταν και η στάση τη προηγούμενη κυβέρνηση και μεταφέρθηκε. Μπορείτε να με διαφωτίσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα το άλλο θέμα. Ε, δηλαδή ε, παρακολουθώ τη χώρα σας ε, και βλέπω ότι επιδεινώνεται η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει εσχάτως εξαφανίστηκε ένας δημοσιογράφος, υπάρχει υπόθεση γονκά αναμένονται τοπικές εκλογές επόμενους μήνες. Ο πρόεδρος γιανουκόβιτς φαίνεται να θέλει τώρα να, εφαρμόσει, να ενισχύσει την ε, θέση του προέδρου, ενώ παλιά που δεν ήταν πρόεδρος ήθελε το αντίθετο. Ε, συνταγματικά πώς θα γίνει. Δεν γίνεται να αλλάζετε τις συνταγματικές ρυθμίσεις κάθε φορά που ε, αλλάζει αυτός που κατέχει την τον προεδρικό θόκο. και επίσης στην Μολδαβία τι θα κάνετε με αυτή την παγωμένη εμπόλεμη ζώνη. Δυστυχώ πρέπει να περιορίσω το χρόνο μιλία σε δύο λεπτά, διότι ο Υφυπουργό πρέπει να φύγει στι 6 και 4 και θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει και στι ερωτήσει. Η κυρία Λούνα Τσέκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω μέλο τη ομάδα των Πρασίνων, ε, εμεί πάντα υποστηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών, ε, την δημοκρατική διαδικασία στην Ουκρανία, περιβαλλοντικέ οργανώσει και ούτω καθεξής. Η βασική μου μέρημνα λοιπόν ε, σήμερα ε, αφορά κάτι που ανέφεραν και κάποιοι συνάδελφοι. Μέλημά μου είναι η μείωση των δημοκρατικών ε, προτύπων της ελευθερίας του τύπου στην Ουκρανία. Το τελευταίο εξάμεινο έχουμε, επιτρέψτε μου τον όρο, κάποια υποδνίδιστα στα γεγονότα. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος εξαφανίστηκε. Ακόμα και ο υπουργό Εσωτερικών είπε ότι μπορεί να είχε σχέση με την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες, ο Βασίλ Κλεμέντιεφ. Ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Μανούκ, ε, ε, ξυλοκοπήθηκε από την αστυνομία. Ε, ο διευθυντής ενό ξένου οργανισμού επίση αγνοεί, συνελήφθη φέτο το καλοκαίρι μία σειρά από γεγονότα, μια ειρηνική διαδήλωση κατά της κατασκευής ενός δρόμου στον Κόρκι Πάρκ στο Κάρκιφ που είναι ε, τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος ε, ε, καταγγέλθηκε ότι υπήρξαν περιστατικά βίας ε, στη διαδήλωση αυτή. Όλα αυτά ανησυχούν όλους μας για το μέλλον της δημοκρατικής διαδικασίας και ε, το πώς μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών στη χώρα σας. Η ερώτησή μου είναι προς τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο, αλλά και προς τον κύριο Κλίμκιν ε, μέλος της κυβέρνησης. Τι κάνετε ώστε να διασφαλίσετε ότι η ελευθερία του συναθρίνεζεσαι, η ελευθερία της γνώμης, η δημοσιογραφική ελευθερία δεν είναι κάτι το οποίο απλώς ε, λέτε στην έκθεση προόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και το υποστηρίζω, αλλά είναι κάτι το οποίο πιστεύετε και κάτι το οποίο είναι εγγυημένο. Ε, κύριε Υπουργέ, εσείς είπατε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ε, θέμα και κατάλληλης νοοτροπίας, αλλά πώς γίνεται, πώς υλοποιείται αυτό στην πράξη. Επίσης, στις 2 Οκτωβρίου θα γίνει μια νέα συνεδρίαση στο Κάρκιφ για το πρόγραμμα του, ε, της Ευρώπης 2012 Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι αυτή η ειρωνική ε, διαδήλωση που θέλουν μια ένα καλό πρόγραμμα για το 2012 θα ε, γίνει πράγματι ειρηνική διαδήλωση. Και τι μπορούμε να κάνουμε για το Euro 2012. Ο κύριος Μπέλντερ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί προσκεκλημένοι από την Ουκρανία, εγώ είμαι Ολλανδός. Και τη Δευτέρα το πρωί ε, είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με ε, Ολλανδικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που ανησυχούν πάρα πολύ ε, για τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ουκρανία, κυρίως στο δυτικό τμήμα, αλλά θέλουν να διευρύνουν τις δραστηριότητε τους και αλλού και ασχολούνται με παιδιά με αναπηρίες σωματικές ή πνευματικές, ασχολούνται με κοινωνικά θέματα και τους ενδιαφέρει η χώρα σας και η κοινωνία σας. Και ε, υπάρχει ε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη χώρα μου. Και εργονιούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι προς τα που ε, πηγαίνει η Ουκρανία πολιτικά. Ανησυχούν μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και ανησυχούν για το κλίμα το πνευματικό και την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία για την κοινωνία, για τα μονομένα άτομα να ε, επιζητούν, ε, να επιδιώκουν τα δικά τους συμφέροντα και η κρατική μηχανή όχι να τους εμποδίζει, να τους βοηθάει στην ολοκλήρωση τους, τους ανθρώπους, να τους υποστηρίζει. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι. Η κόρη μου ίδια το καλοκαίρι, ε, δύο εβδομάδες στο Κάρχιβ, ε, κατά τη διάρκεια των διακοπών της έκανε μαθήματα αγγλικών και γύρισε κατεθουσιασμένη. δίδασκε αγγλικά δηλαδή. Ε, εμείς βλέπουμε και θέλουμε να έχει μια θέση η Ουκρανία στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε και μια Ουκρανία που να υποστηρίζει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες στην κοινωνία κτλ. Με δύο λόγια, θέλω να απευθύνω μια έκκληση. Πραγματικά διασκεδάστε αυτούς τους φόβους, διαλύστε αυτές τις αγωνίες ε, για ε, το κλίμα αυτό που είναι, φαίνεται αρνητικό και οι άνθρωποι είναι σφιγμένοι και ως προς τις ελευθερίες. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Πέτρελ. <clears throat> Ήμουνα στην Ουκρανία πριν μετά από τις εκλογές ε, με το ρόλο του παρατηρητή και διαπίστωσα κάτι ιδιαίτερο. Συνάντησα κάποιους φοιτητές οι οποίοι ε, μέσα στην ίδια μέρα ε, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον ένα υποψήφιο και μετά άλλαξαν γνώμη και υποστήριξαν τον άλλον. Και τους ρώτησα ποιον θα ψηφίσετε και μου είπανε κανέναν. Γιατί δεν μας ε, ε, ε εκπροσωπεί κανένα ουσιαστικά. Αυτό είναι ένδειξη απάθειας από πλευράς των νέων. Με χαροποιεί λοιπόν το γεγονός ότι σήμερα βλέπω ότι υπάρχει κάποια σύγκληση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δυσκολίες ε, και διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά αν υπάρχει πολιτική συνένεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ε, σε θέματα ε, ευρωπαϊκών ε, προτύπων, όπως για παράδειγμα την κοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη σχέση μεταξύ πολιτών και κράτους. Ε, αυτή η συνένεση θα μπορέσει να μειώσει αυτή την απάθεια την οποία έχουν αυτή τη στιγμή οι, Ευρωπαίοι, οι Ουκρανοί ψηφοφόροι, κυρίως οι νέοι. Επίσης, να σας πω ότι όταν η χώρα μου ετοιμαζόταν για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωρήσαμε καλά διότι μπορέσαμε να έχουμε μια ευρεία πολιτική συνένεση για τα όσα θεωρούσαμε ότι θα είχαν σημασία και θα είχαν προωθήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Σλοβενία. Ε, συνειδητοποίησαμε όλοι τι σήμαινε η ένταξη της Ευρωπαϊκής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα πρέπει το ίδιο να κάνει και η χώρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πέτερλε. Στη συνέχεια για δύο λεπτά ο κύριος λίδη και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Τάραζουκ. Θα διαπιστώσετε και οι δύο σώμασοι πόσοι ε, εξημών είναι φίλοι της Ουκρανίας. Έχουμε συζητηθεί και στο παρελθόν, αλλά ο Μπόρις μπορεί να σας επιβεβαιώσει ότι εγώ είμαι φίλος της Ουκρανίας. Γι' αυτό μην εκλάβετε αυτά που θα σας πω ως επίκριση, αλλά ως ανησυχία για την Ουκρανία. Καταρχάς, η Συμφωνία Διασύνδεσης και η Συμφωνία Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου και οι διαπραγματεύσεις ε, για τη Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για το πρόοδο που έχει καταφέρει να επιτύχει η Ουκρανία. Υπάρχουν ανησυχίες από πλευράς Βερξελών. Εσείς κύριε Υπουργέ, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόσκομα από πλευράς Ουκρανίας για να επιτευχθούν όλα τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Δεύτερον, συζητήσαμε και πολιτική γνωρίζετε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονται τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν είναι και το πιο σημαντικό θέμα μεν στον κόσμο, αλλά γνωρίζετε ότι μας ανησυχεί ε, η δημοκρατική διαδικασία στην Ουκρανία. Εδώ και χρόνια λέω στον Μπόρις ότι κάποιοι από τους εκλογικούς νόμους στην Ουκρανία είναι μάλλον περίεργοι δεν θα σας κάνω εγώ διάλεξη τώρα, αλλά μήπως θα μπορούσατε να επανεξετάσετε τους εκλογικούς νόμους σας και να δείτε τι ε, εκλογικούς νόμους έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γεωργία αυτή τη στιγμή αλλάζει το σύνταγμά της και χρησιμοποιεί ως πρότυπο το πολωνικό σύνταγμα. Το ξέρω ότι έχετε υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία για την παράταση του γιατί, των βάσεων. Ε, πιστεύετε ότι οι βάσεις οι ρωσικές θα είναι καλές για την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ τον κύριο Λίζεκ. Ε, λυπάμαι, έχετε πολύ λίγο χρόνο για να απαντήσετε γιατί δυστυχώς πρέπει να φύγετε σε λίγο. Δεν μπορέσαμε να περιορίσουμε τις παρεμβάσεις μας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, το αφήνω σε εσά. Αν μείνετε ίσως λίγο παραπάνω, να, θα μπορέσετε να απαντήσετε. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Uh, firstly, uh, ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις και για τις ανησυχίες και τα μελήματά σας. Βεβαίως, καταλαβαίνω τι εννοείτε. Δεν είμαι σε θέση μάλλον να μπω σε λεπτομέρειες για όλα τα ζητήματα ε, που ε, θέσατε. Θα προσπαθήσω όμως, αν μη τι άλλο, να απαντήσω κάποια βασικά σημεία με βασικά μηνύματα. Πρώτον, για την κατάργηση της θεώρησης διαβατηρίων. Το θέμα είναι πολιτικό και τεχνικό. Ήδη σας είπα ότι είμαι μέγας υποστηρικτής. Πώς να το πω. Ε, του να απαλλάξουμε τη συζήτηση αυτή από το πολιτικό της ε, φορτίο και να ε, συζητούμε μόνο τα τεχνικά ζητήματα. Βεβαίως, κάνει προσπάθειες και αλλαγές και δεν είναι μόνο νομοθετικές, είναι και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ε, στην Ουκρανία που πρέπει να γίνουν και εφαρμογή. Θα σας δώσω με μεγάλο ενδιαφέρον, αν σας ενδιαφέρει, ένα τέτοιο κατάλογο και μπορεί να είναι και χρήσιμο. Το δεύτερο που είπε ο Πάβελ Κόβαλ με ανησύχησε λίγο, διότι δεν βλέπω πουθενά ε, σημεία που να ε, χρειάζεται να σας προκαλούν ανησυχία ε, για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Ταρασούπ είπε ότι εδώ έχουμε εθνική συνένεση. Ε, η πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είναι ε, μόνο ένα πλαίσιο αλλά και μια κατεύθυνση, ένας μπούσουλας, μια πηξίδα για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα, για την πιθανή τελωνιακή ένωση με τη Ρωσία ε, που έχει δημιουργήσει η Ρωσία με το Καζακστάν και τη Λευκορωσία. Αν αφήσουμε την πολιτική στην άκρη, πώς θα μπορούσαμε και θεωρητικά έστω να το κάνουμε, γιατί θα πρέπει να ε, επαναδιαπραγματευτούμε τις υποχρεώσεις και τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους ενταχθήκαμε στον ΠΟΕ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ε, στον ΠΟΕ ποτέ είναι πρωτοφανές, δηλαδή και από ρεαλιστικής πλευράς και από ε, πολιτικής. Ο πρόεδρος μας το έχει επαναλάβει πολλές φορές και το έχει τονίσει ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να ενταχθούμε στην Τελωνιακή Ένωση με τη Ρωσία. Και μεταξύ άλλων γιατί έχουμε κάποιες υποχρεώσεις από τον ΠΟΕ αλλά και άλλα ζητήματα που μας δεσμεύουν. Άλλο σημείο, αυτό που αφορά το Μαυροβούνιο. Θα μπορούσα να το συζητήσω σε λεπτομέρειες, αν θέλετε, να το συζητήσουμε και σε λεπτομέρειες. Αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις μας είναι η πρόσβαση στην αγορά ε, χάλιβα ε, του Μαυροβουνίου, γιατί έχει αυξήσει σημαντικά ε, τους δασμούς για προϊόντα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία, ιδιαίτερα τρόφιμα. Εμείς σεβόμαστε πλήρως ε, την πορεία του Μαυροβουνίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το ίδιο με μας, αλλά δεν μπορούμε να ε, δεχτούμε ότι μας αυξάνουν τους δασμούς και τους διπλασιάζουν. Ε, ή ας πούμε την πρόσβαση Δεν ξέρω αν έχει να κάνει αυτό και με τη Σερβία. Θέλετε να το συζητήσουμε ευρύτερα ε, και σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Ναι, παρακαλώ. Ναι, μπορώ να σας δώσω και γραπτή ενημέρωση αν σας ενδιαφέρει, γιατί υπάρχει, για την υπερθνιστερία. Εμείς είμαστε πλήρως προσυρωμένοι στην επίλυση αυτής της σύγκρουσης και Υπάρχει ένα σύστημα διαπραγματεύσεων 5 συν 2 και είμαστε υπέρ της πλήρους ανανέωσης ε, των συνομιλιών και θα μπορούσαμε εδώ ακριβώς να βοηθήσουμε να εξελιχθούν τα πράγματα προς την καλή κατεύθυνση. Για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2012 είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο και είμαι πεπισμένος ότι αυτό το θέμα δεν είναι σε καμία περίπτωση ε, θέμα κύρους ή προετοιμάσεων, είναι θέμα εθνικής υπερηφάνειας. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι σχεδόν θρησκεία στην Ουκρανία. Και καταλαβαίνουμε ότι αν δεν επιτύχουμε εκεί θα είναι καταστροφή και για την Ουκρανία και για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερο πρωτάθλημα μαζί με τους Πολωνούς μας φίλους που τόσο διοργανώνουμε. Ε, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε αντίστοιχη υπηρεσία γραφείο καταπολέμησης διαφθοράς. Χρειάζεται και ένα νομοθετικό πλαίσιο και ε, μπορώ να σας ενημερώσω και πάλι γραπτός για τα πρακτικά βήματα ε, σε αυτή την κατεύθυνση. Η ε, Επίτροπος κυρία Άστον έκανε κάποια τέτοια παρατήρηση και σχόλια. Θα τα μελετήσουμε στενότερα. Εγώ δεν το είδα. Δεν είχα την ευκαιρία να το μελετήσω. Απλώς το άκουσα. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση δεν έχει καμία σχέση με συνεργασία στρατηγική, ειδικέ σχέσεις με την Ουκρανία η λύση. Αυτό που ενδιαφέρει την Ουκρανία είναι η πλήρης ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μελλοντικά. Ένταξη και καμία άλλη μορφή συνεργασίας. Θα δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε, πώς προετοιμαζόμαστε, πώς διαμορφώνουμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι τώρα στο θέμα στα θέματα που σας ανησυχούν για τις περιφερειακές δημοτικές εκλογές. Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι ουδής τέλειος εδώ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ε, έγιναν κάποιες αλλαγές τους νόμους που διέπουν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ε, αυτό είναι το θέμα. Θα πρέπει να δείτε την κατάσταση πιο συνολικά. Ερώτηση. Γιατί κάποια πολιτικά ε, κόμματα που υπάρχουν εδώ και χρόνια, γιατί δεν έχουν καταγράψει, δεν έχουν δηλώσει τα τοπικά τους παραρτήματα. Η απάντηση συνεπής και συνολική θα ήταν ε, ο νέος εκλογικός νόμος, εκλογικός κώδικας ε, και υπάρχει πρόθεση και πολιτική δέσμευση να γίνει αυτό στο Κοινοβούλιο. για τη διαφάνεια και τους παρατηρητές από διεθνεί οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να είναι ανοιχτέ οι εκλογές. Ελάτε να, δείτε τις εκλογές και πώς θα γίνουν γιατί οι ελεύθερες εκλογές και οι δίκες εκλογές είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ την Ουκρανία. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να καλύψω όλα τα θέματα που με ρωτήσατε, αλλά είμαι πρόθυμος να σας στείλω και γραπτές απαντήσεις στο βαθμό που το επιθυμείτε για αυτά τα θέματα. Για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, αυτό ίσως χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι ε, για τις ερωτήσεις σας. Και ευχαριστώ τον ε, κύριο Υπουργό. Κύριε Τάραζουκ, έχετε κάποια λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε εσά. Παρακαλώ. Uh, well, ε, ευχαριστώ. Ε, ε μας απίθυναν ερωτήσεις προς τον κύριο Κλίμπκιν και προς εμένα, τα μέλη της Επιτροπής, ε, αρκετές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου, προσπαθούσα να ξεχάσω ότι είμαι μέλος αντιπολίτευσης στην Ουκρανία. Ε, προσπαθούσα να εστιάσω στα βασικότερα ζητήματα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι ζήτησα να μοιραστεί του να, να, ε, οι ηγέτες όλων των αντιπολιτευτικών κομμάτων της ε, Ουκρανίας ε, να απευθύνουν έκκληση στην Επιτροπή μας και εξάλλου έχουμε στείλει και επιστολή στον κύριο Φανναρόμπα και στον πρόεδρο Μπαρόσο και στον πρόεδρο Μπούσεκ και προς όλους σας όλους εσάς, αξιότιμα μέλη του, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, για τις επικείμενες ε, εκλογές ε, στη, στη, την 31η Οκτωβρίου. Γιατί έχει περάσει ένας αντιδημοκρατικός ε, νόμος και υπάρχει συστημική δυνατότητα ευρείας νοθείας και απάτης. Εφτά συστημικά προβλήματα υπάρχουν. Εμείς η Ηνωμένη Αντιπολίτευση της Ουκρανίας τα έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα και θα ήθελα ε, να σας θυμίσω ότι η Ηνωμένη Αντιπολίτευση έχει απευθύνει η μαζική έκκληση κατά αυτού του νόμου. Άκουσα ανησυχίε από διακεκριμένους βουλευτές του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Και όπως και κάποιοι από εσά, έτσι και εμείς στην αντιπολίτευση στην Ουκρανία ανησυχούμε γιατί οι αρχές αποκλίνουν από τις ευρωπαϊκές αρχές, αποκλίνουν από την δημοκρατική πρόοδο που επιτύχαμε μετά τη νίκη της δημοκρατίας στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Πορτοκαλή Επανάστασης. Δεν μπορώ παρά να αναφερθώ και στην ε, αξιολόγηση, στη πληρέστατη ε, αξιολόγηση που έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου ενός ε, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ε, δεν μιλάμε μόνο για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Υπάρχουν ε, παραβιάσεις των βασικών δικαιωμάτων, ε, παραβίαση της ελευθεροτυπίας, ε, της ελευθερίας έκφρασης και μην ξεχνάτε ότι στην, σε μια άλλη μελέτη που συγκρίνει τις κοινοβουλευτικές επιδόσεις των χωρών εκφράζεται ανησυχία για την υπαναχώρηση από την πρόοδο που είχε σημειωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια στην πορεία εκδημοκρατισμού της χώρας. Υπάρχουν πολύ σοβαρέ ε, ανησυχίε λοιπόν στην αντιπολίτευση και σας παραπέμπω σε αυτή την επιστολή που στείλαμε. Θα ήθελα δε να κάνω και ένα σύντομο σχόλιο για τις ε, δυνάμεις ασφαλείας και τον κύριο Χοροσκόφσκι που είναι επικεφαλής ε, είναι μεγιστάνας ε, των ε, μέσων μας ενημέρωση επικεφαλής μυστικής υπηρεσίας, ε, μέλος του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου που μπορεί να αποπέμπει και να διορίζει τους δικαστές. Προφανέστατη δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων εφόσον συγκεντρώνονται σε αυτές οι ιδιότητε σε ένα άτομο. Ε, και τους τελευταίους μήνες ε, η υπηρεσία πληροφοριών, η μυστική υπηρεσία ε, επιτίθεται στην, σε μέλη της αντιπολίτευσης και πλαστοποιεί αποδεικτικά στοιχεία σε διάφορες ποινικέ διώξεις. Αυτά, αυτά κάνουν στην Ουκρανία. Είναι όπως η, η KGB, η KGB στην Σοβιετική Ένωση δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε πραγματική ανησυχία για την απόπειρα της τωρινής κυβέρνησης ε, να ε, παρεμβαίνει στα ισοτοκομματικά, παραδείγματος χάρη. Ε, Όπω το πάρτι τη ε, Γιούλια Τιμοσέγκο, που είναι το μεγαλύτερο, Τζούλια Τιμοσέγκο, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα τη αντιπολίτευση, Ε, και ε, ορισμένες φορές ε, παρουσιάζουν υποψηφίους σαν να είναι δικοί τους. Δηλαδή κάνουν και απίστευτα πράγματα πλέον τη διάρκεια της δημοκρατικής διαδικασίας, για τις εκλογές δηλαδή. Ελπίζω τελικά να ε, ε, καταλήξουν διαπραγματεύσεις για την Τελωνιακή Ένωση με τη Ρωσία. Η Βαρόνια στον ε, εκφράστηκε όπως είπατε και εξεπλάγην κι εγώ. Παρά αυτά που είπε, παρόλα αυτά που είπε το γραφείο τύπου του Κοινοβουλίου, αυτά έγιναν. Θυμηθείτε περίφημες δηλώσεις από έναν ε, άλλο υψηλό βαθμό αξιωματούχο της Ένωσης, ε, τον κύριο Φερχόιγγεν. Συγγνώμη, αλλά είναι αρνητικές αυτές οι τάσεις ε, που παρατηρούνται και ελπίζω ότι εσείς θα κάνετε την αξιολόγησή σας εγώ είμαι, είπα, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την προσχώρηση της Ουκρανίας στην Ένωση και με αυτή την ιδιότητα θα ήθελα να ε, σας πω ότι θα ζητώ διευκρινιστική δήλωση από πλευράς της ΥΠΑ της εκπροσώπου στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, από πλευράς δηλαδή της Βαρόνης Άστον για να εξηγήσει τι εννοούσε με αυτή τη δήλωση. Ε, τέλος, ε, για την υπεράσπιση της ελευθεροτυπίας ε, και των δημοσιογράφων που εκφοβίζονται και φύστανται ξυλοδαρμούς, τι κάνετε, τι κάνουμε, να σας εξηγήσουμε πρόσφατα. Η αντιπολίτευση συμφώνησε ότι η Επιτροπή Ελευθεροτυπίας ε, θα έχει ως πρόεδρο έναν ε, δημοσιογράφο, τον Αντρέη Σιψέγκο, που είναι από ε, τους προτεργάτες στο κίνημα της υπεράσπισης ελευθεροτυπίας. Ε, και είναι από τα βασικά κόμματα τη αντιπολίτευση, θα έχουμε μεγαλύτερη μόχλευση. Αλλά μην ξεχνάτε, αντιπολίτευση είμαστε. Δεν έχουμε ε, αρκετέ ε, ψήφου για να παρεμποδίσουμε εμεί σε μια νομοθετική διαδικασία για να εμποδίσουμε αυτέ τι εξελίξει στην Ουκρανία. Τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό, υπάρχει συμφωνία με τη Ρωσία για την παραμονή της ναυτικής βάσης στον Εύξηνο Πόντο στις διαπραγματεύσεις ε, με τη Ρωσία ε, ε, συμμετείχε ένα μέλος της αντιπολίτευσης που με διαβεβαίωσε ότι απειλείται η σταθερότητα και η ασφάλεια της Ουκρανίας όσο παραμένει ο ρωσικός στόλος στον εύξηνο πόντο. Ελπίζω να ε, μην γίνει αυτό το λάθος, να μην παραβιαστεί έτσι το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας. Ε, είμαι σίγουρος ότι ε, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, δηλαδή άλλου είδους μοχλεύσεις, πιέσεις που μπορούν να ασκηθούν, χάρη στις οποίες όταν εμείς ανέβουμε στην εξουσία να μπορέσουμε να καταγγείλουμε τη συμφωνία με τη Ρωσία. με, αυτά τα πρόσχαρα θα τελειώσω και θα σας πω, Πρόεδρε, και στα όλα τα μέλη της Επιτροπής που ήταν αρκετά υπομονετικά ώστε να μείνουν μέχρι τέλους. Ε, να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη χώρα μου και για την ε, επέκταση της ε, δημοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους σας. Τα τελευταία σας λόγια φυσικά μας βρίσκουν και εμάς σύμφωνους ε, και εμείς ε, αυτό θέλουμε και προσπαθούμε να το επιτύχουμε. Επόμενη συνεδρία της Επιτροπής 5 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί στις Βρυξέλλες. Ε, πέρασε συνεδρία σας. Καλό σας βράδυ.